Liebe Kollegen, meine Damen und Herren, äh, ich möchte die heutige Sitzung. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κηρύξω την έναρξη τη ειδική επιτροπή. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε σε όλες τις γλώσσες του Κοινοβουλίου και καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω αν έχετε παρατηρήσει σχετικά με την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, οπότε εγκρίνεται. Δεν έχω να σας κάνω ιδιαίτερες ε, ε, προτάσεις τάσεις ή ανακοινώσεις οπότε πάμε στο τρίτο σημείο έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης ε, έχετε από αυτού κάτι ε, τότε εγκρίνονται και τα πρακτικά και ερχόμαστε τώρα στο σημερινό μας πρόγραμμα καταρχήν είναι μεγάλη χαρά για μένα να ε, καλωσορίσω εδώ τον Τομάσο Παντοσόπα ο οποίος σε πολλά σημεία έχει συμβάλει εις ε, την συγγραφή και στη διαμόρφωση της ευρωπαϊκής ιστορίας. Ως εκ τούτου δεν ε, χρειάζεται να σας πω λεπτομέρειες από το βιογραφικό του, αλλά ξέρετε ότι είναι μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, του Ελεκτρικού, ε, ε, ε Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρόεδρος του Ιδρύματος για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα από το 2005-2006 και όπως ξέρετε ε, θα ε, παρουσιάσει ε, τώρα το θέμα αυτό που είχε που αναφέρεται εις το Ίδρυμα Νότρο Ροπ το οποίο είχε ιδρύσει ο Ζακ Ντελόρ. Θα ήθελα επίσης να σας πω ότι υπάρχει παρουσίαση της, της συνεδριάσεως στο διαδίκτυο. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή που με κάλεσε αυτή η Επιτροπή στην ακρόαση αυτή διότι ε, εδώ ε, έχετε σαν στόχο να εξετάσετε τα θέματα της κρίσεως συνολικά. Διότι όντως η κρίση αυτή αναφέρεται σε τόσους τομείς που συγκροτούν τις ε, εντολές ε, των διαφόρων επιτροπών ώστε χωρίς να υπάρχει μία ειδική ε, επιτροπή για την κρίση θα ήταν κατακαιρματισμένη η αντιμετώπιση των θεμάτων και θα εμπόδιζε να συλλάβουμε όλες τις απόψεις της κρίσεως αυτής. Το σημερινό πρόγραμμα Αναφέρεται στην ε, ε, ε, παγκόσμιο διακυβέρνηση και ε, θα αναφερθώ στο συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα χωρίς ε, να αναφερθώ στις γενικότερες ε, σκοπιές της κρίσεως και θα ήθελα καταρχήν να κάνω μία εισαγωγή για την θέση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην κρίση αυτή. Δεύτερον, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα του εάν η κρίση έχει καθοριστεί από την παγκοσμιοποίηση, εάν η παγκοσμιοποίηση είναι η αιτία της κρίσης δηλαδή. Το τρίτο μου θέμα θα είναι ποια είναι τα μέσα για να να διορθώσουμε την κατάσταση, δηλαδή πώς μπορεί να διαμορφωθεί η παγκόσμιος διακυβέρνηση για να αποφευθεί η επανάληψη μιας τέτοιας κρίσης και τέταρτον τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να συμβάλλει εις ε, την ε, αναθεώρηση της ε, παγκοσμιοποιημένης διακυβέρνησης. Η πρώτη μου λοιπόν παρατήρηση συνοψίζεται στην εξής δήλωση η κρίση δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να είναι το πρώτο θύμα της κρίσεως αυτής. Γιατί δεν προέρχεται δηλαδή η κρίση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν προέρχεται διότι οι ε, παράγοντες κλειδιά οι οποίοι κρύβονται πίσω από την κρίση αυτή ήταν πολύ πιο τονισμένοι και επηρέασαν πολύ περισσότερο άλλες περιοχές της Ιφιλίου πέραν της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Παραδείγματος χάρη η ε, ακραία φονταμενταλιστική ιδεολογία της αγοράς ε, που έλεγε ότι πάντοτε οι αγορές έχουν δίκιο και οι οικονομικές αγορές ε, κινούνται πάντοτε προς μία ισορροπία ότι ο βασικός ρόλος, ρόλος του κυβερνήσεως είναι να μειώσει το μέγεθός του και να συρρυκνωθεί για να αφήσει ε, την, ε, ε, τις αγορές να λειτουργήσουν. Αυτές οι φονταμενταλιστικές απόψεις ήταν πολύ πιο ενισχυμένες στην Ευρώπη από ό,τι σε άλλες ε, περιοχές της Ιφιλίου. Επίσης η ιδέα ότι η διεθνής ολοκλήρωση μπορεί να γίνει χωρίς κάποια δημόσια δομή είναι το αντίθετο από τον τρόπο με τον οποίο έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή η ακολουθήθηκε μία μορφή που δεν ε, ε, επηρεάζεται από τις ε, αρχές ενώ εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει κοινοβούλιο, υπάρχει νομική αρχή, υπάρχει προϋπολογισμός, υπάρχουν δηλαδή όλα τα στοιχεία τα οποία συμπληρώνουν τους μηχανισμούς της αγοράς. Οπότε η ισορροπία μεταξύ ε, της αγοράς και της δημοσίας πλευράς ε, υπάρχει στο παγκοσμιοποιημένο υπάρχει στην Ευρώπη και γι' αυτό ε, δεν επηρεάζεται τόσο όσο η σκηνή της παγκοσμιοποίησης. Επίσης, ε, μία από τις στάσεις οι οποίες είναι στη βάση αυτής της κρίσεως είναι και πάλι λιγότερο τονισμένη. Δηλαδή η Ευρώπη έχει διαμορφωθεί διαφορετικά. και όχι ε, στο ίδιο επίπεδο όσο άλλες οικονομίες. Τέλος, οι ανισορροπίες που ήταν τόσο τεράστιες στην Αμερική, ε, το εμπορικό, το εμπορικό έλλειμμα, το φορολογικό έλλειμμα ε, της Αμερικής δεν αντικατοπτρίζονται στον ίδιο βαθμό στην Ευρώπη. Οπότε οι περισσότεροι παράγοντες που συνέβαλαν στην Κρήτη δεν ήταν χαρακτηριστικά ευρωπαϊκά στοιχεία και αν ο υπόλοιπος κόσμος είχε ακολουθήσει τα χαρακτηριστικά της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να μην είχε υπάρξει αυτή η κρίση. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να είναι το πρώτο θύμα της κρίσης διότι την έπληξε η, η κρίση, μάλλον την συνέλαβε εξαπίνης σε κάποια στιγμή ατελούς οικοδομήσεως που την κατέστησε πολύ πιο ευάλωτη από ό,τι άλλες πλευρές του κόσμου. Δηλαδή δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση η διαχειριστική δυνατότητα, υπάρχει στο, επίπεδο των κρατών αλλά προφανώς στο επίπεδο των κρατών παίρνει ένα χαρακτήρα στηρίξεως και προστασίας της ε, εθνικής οικονομίας και όχι τόσο πολύ της παγκοσμίου οικονομίας μάλλον της ευρωπαϊκής οικονομίας και γι' αυτό είδατε ότι εάν χρειαστεί να βοηθήσει κανείς τράπεζες οι τράπεζες αυτές βασίστηκαν σε εθνικά εργαλεία και αυτό δημιούργησε και σοβαρές τριβές σε ορισμένες χώρες όταν οι τράπεζες που αντιμετώπιζαν προβλήματα ήταν πολυεθνικές το ίδιο είδαμε και στις βιομηχανίες όπως η αυτοκινητοβιομηχανία και τέλος και επίσης επίσης πολύ σημαντικό, το βλέπουμε τώρα όταν μία χώρα πλέον είναι υποποίηση και όχι ένας μεμονωμένος τομέας ή μία τράπεζα. Εδώ μιλάμε για την ελληνική κρίση. Η κρίση λοιπόν αυτή δεν προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να είναι το πιο σοβαρό θύμα. Ε, η αιτία της ε, κρίσεως και η παγκοσμιοποίηση. Δεν νομίζω ότι η παγκοσμιοποίηση ευθύνεται για την κρίση, αλλά ορισμένε ε, πτυχές της παγκοσμιοποίησης έχουν διευκολύνει μία μακρά παράταση μίας απαράδεκτης ε, κατάστασης γεγονότων και όταν έφτασε ο κόμπος στο χτένι τότε αυτό έγινε πάρα πολύ θεαματικά. Δηλαδή τα πράγματα είχαν ήδη επιδεινωθεί πάρα πολύ ενώ εάν είχε υπάρξει κάποια ένδειξη πιο νωρίς ενδέχεται η, η κρίση αυτή να μην ήταν τόσο σοβαρή να μην ήταν μια κρίση αλλά μια φυσιολογική προσαρμογή στην ε, οικονομία όπως συμβαίνουν ανα πάσα στιγμή. Ποιες είναι οι επιπτώσεις της παγκοσμιοποίησης που διευκόλυναν την κρίση. Καταρχήν είναι η θέση του αμερικανικού δολαρίου. Δηλαδή μία χώρα με τεράστιο έλλειμμα ήταν η χώρα η οποία είχε εκδώσει το διεθνές νόμισμα και ε, αυτό ε, κατέστησε το, ε, τη δυνατότητα να συσσωρευτεί αυτό το έλλειμμα πολύ εύκολη και δεν προχώρησε η εξέλιξη όπως θα είχε είχε συμβεί σε μια χώρα άλλη όπου θα υπήρχε μια ανεπάρκεια πόρων, δεν θα υπήρχε δυνατότητα να εξυπηρετήσει η χώρα αυτή τα δάνειά της και όταν η ελληματική χώρα βέβαια εκδίδει το νόμισμα της υφηλίου δεν υφίσταται τα ίδια στοιχεία πειθαρχία τα οποία υφίστανται οι άλλες χώρες. Υπάρχει όμως και μία άλλη άποψη της παγκοσμιοποίησης που είναι το γεγονός ότι η πολύ υψηλή ρευστότητα η οποία επέτρεψε την ε, ανάπτυξη ε, της ε, φούσκας στον οικοδομικό τομέα στις Ηνωμένε Πολιτείε θα είχε δημιουργήσει μία έξαρση πληθωριστική όπως συνήθως συμβαίνει όταν ε, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη δημιουργία χρήματος επί πολύ μακρύ χρονικό διάστημα. Πλην όμως ε, υπήρχε μία καταστολή ε, των πληθωριστικών πιέσεων με την εισαγωγή φθηνών εισαγωγικών αγαθών από άλλες χώρες όπως η Ασία. Οπότε δεν παρήχθησαν τα φυσιολογικά ε, οι φυσιολογικές επιπτώσεις ούτε εσωτερικά σαν πληθωριστικές πιέσεις διότι ε, υπήρχε η δυνατότητα προσβάσεως σε φθηνά μεταποιημένα αγαθά που διατήρησε σταθερές τις τιμές ούτε διεθνώς όπου η ε, πρόκληση ενός μηχανισμού πειθαρχίας ο οποίος λειτουργεί για χώρες οι οποίες ε, ε, δεν εκδίδουν το ε, νόμισμα απόθεμα θα είχε ισχύσει. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η παγκοσμιοποίηση δημιουργεί προβλήματα και ως εκ τούτου είναι κάτι το κακό. Αλλά ορισμένες πτυχές του τρόπου με τον οποίο η παγκοσμιοποίηση εξελίχθηκε κατά την τελευταία 20 ετία έχει δημιουργήσει μία παράταση των ε, ανισορροπιών οι οποίες ε, κάποια στιγμή δεν θα μπορούσαν να διορθωθούν παρά μόνο με μία κρίση. Αυτό δεν είναι όμως ενάντια της παγκοσμιοποίησης, είναι ενάντια μίας παγκοσμιοποίησης η οποία στερείται στοιχείων παγκοσμίου διακυβέρνησης που είναι και το θέμα αυτής της συνεδριάσεως που ε, εμποδίζει να υπάρξει ενσωμάτωση των αγορών με ε, κοινέ ε, γενικές πολιτικές ιδίως από πλευράς μακροοικονομικής πειθαρχίας και νομισματοχής τάξεως. Ποια είναι τώρα ε, η λύση, πώς μπορεί να αναθεωρηθεί η διακυβέρνηση αυτή. Η κρίση ήδη έχει προκαλέσει μία υγιή ε, αναμόρφωση, οδήγησε στις DG7 να μετατραπούν σε G20 όπου συμμετέχουν περισσότερες χώρες. Αυτή η κίνηση είναι ε, θετική διότι η G7 δεν ήταν ε, αντιπροσωπευτική της Ιφιλίου δεν ε, ε, εκπροσωπώντουσαν οι χώρες που είχαν τα μεγαλύτερα πλονάσματα δεν μπορούσαν να υπάρξουν ουσιαστικές εμπορικές συζητήσεις διότι καλύπτονται μόνο μερικές από τις ε, χώρες, δηλαδή οι βιομηχανοποιημένες χώρες, ενώ η G20 που υπάρχει τώρα ε, αντιπροσωπεύει πολύ καλύτερα την παγκόσμια οικονομία. Συγχρόνως η διεθνή συνεργασία η οποία βαθέζεται, βασίζεται στα G, δηλαδή στα groups, στις ομάδες, είτε τα G7, τα G20 ή τα G2 όπως λένε ορισμένοι, <clears throat> κατά τη γνώμη μου, εμποδίζει να υπάρξει μία διεθνή συνεργασία που θα περιλαμβάνει τα θεσμικά στοιχεία τα οποία είναι στο επίκεντρο των διεθνών οργανισμών που δημιουργήθηκαν μετά από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, τα Ηνωμένα Έθνη και ο ΠΟΕ. Όταν απουσιάζουν αυτοί οι οργανισμοί και υπάρχουν απλώς επιτροπές χωρίς ένα θεσμικό όργανο το οποίο να αντιπροσωπεύει ολόκληρο τον κόσμο και να εξασφαλίζει τη διακυβέρνηση μεταξύ των συναντήσεων ε, και να αναλύει τα βασικά θέματα δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο καλό αποτέλεσμα διότι δεν υπάρχει ένα σημείο όπου να λαμβάνονται αποφάσεις προς το γενικό συμφέρον. Ένα λοιπόν από τα βασικά στοιχεία για την ε, αναμόρφωση της ε, παγκοσμίου διακυβερνήσεως θα ήταν να επαναφερθούν ε, τα σημεία διεθνής συνεργασίας όχι σε συνελεύσεις αλλά να επανέλθουν σε θεσμικά όργανα που θα έχουν μία διοίκηση και θα επιτρέψουν να εκπροσωπείται η ραχοκοκαλιά της παγκοσμίου διακυβέρνησης. Επίσης κάτι το οποίο δεν έχει ληφθεί υπόψη επαρκώς στη συζήτηση για τις ε, μεταρρυθμίσεις είναι η αναθεώρηση της διεθνούς νομισματικής τάξεως. Έχουν υπάρξει ε, πολλά σχόλια, πολλές χώρες οι οποίες ζητούν μια τέτοια μεταρρύθμιση διότι τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα είναι απλώς ε, εργαλεία με τα οποία διάφορες ε, δομές ε, ε, διεθνών νομισματικών σχέσεων μπορούν να επιτρέψουν να υπάρχει μία πιο σταθερή έκφραση από ότι το καλάθι είναι ένα εργαλείο όπου όμως θα έπρεπε να υπάρχει και η τιμή των πρώτων υλών που να συνυπολογίζεται υπάρχουν ήδη διάφορα στοιχεία του διεθνούς νομισματικού νομισματικού συστήματος και κατά τη γνώμη μου το θέμα ε, μίας διεθνούς νομισματικής μεταρρύθμισης είναι ε, απαραίτητο να συζητηθεί εάν μπορεί να παραμείνει μία τέτοια τάξη. Τέλος, βλέπω ότι τελειώνει ο χρόνος μου, τι θα μπορούσε να κάνει από αυτού η Ευρώπη. Νομίζω ότι ξεκινάμε από εκεί που, από αυτά που σας είπα. Δηλαδή ε, ε, πρέπει σε περιφερειακό επίπεδο να δημιουργήσει μία τελείως διαφορετική, έχει δημιουργήσει μία τελείως διαφορετική ολοκλήρωση διεθνή από ό,τι στα άλλα μέρη του κόσμου. Υπάρχει νομοθετική αρχή, σύστημα, δεν υπάρχει μόνο η αγορά αλλά υπάρχει και η πλευρά της ε, δημοσίας αρχής μιας ολοκληρωμένης οικονομίας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περαιτέρω σε περιορισμένο βαθμό δεχτεί το βασικό στοιχείο χωρίς το οποίο δεν υπάρχει αποτελεσματική διακυβέρνηση δηλαδή η δυνατότητα να ληφθούν αποφάσεις ακόμη και αν ε, ε, οι συμβαλόμενοι γύρω από το τραπέζι διαφωνούν. Μπορεί να υπάρξει η Ευρωπαϊκή, ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία δυνατότητα για πολιοψηφική απόφαση η οποία δεν υπάρχει πλέον στην παγκόσμια σκηνή. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παρουσιάσει ένα πρότυπο για καλύτερη ε, παγκόσμιο διακυβέρνηση και να το εφαρμόσει πιο συνεπώς και επανέρχομαι στο σημείο από το οποίο ξεκίνησα. Δηλαδή ενδέχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι το πρώτο θύμα της κρίσεως διότι είναι ε, ατελής ένωση και μία ατελής ένωση μπορεί να επιβιώσει σε κανονικές εποχές αλλά εκτίθεται σε μεγάλους κινδύνους σε περίπτωση τέτοιας κρίσεως. Ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε τώρα να ακούσουμε τις ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Θα δώσω χρόνο να μιλείτε για απαντήσεις. Θα αρχίσω με τους συντηρητικούς. Ποιος θέλει να θέσει πρώτος ερωτήσεις. Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για την ομιλία σας και θα ήθελα να σας ε, ευχαριστήσω ε, ότι, διότι ήσασταν διαθέσιμος και στις επιτροπές οι οποίες ενεπλάκησαν σε αυτή την εκδήλωση. Ε, σήμερα Λέγεται συνεχώς ότι οι αρχηγοί των κυβερνήσεων για να επιλύσουν ε, το πρόβλημα της Ελλάδος ε, προωθούν ένα συνδυασμένο σύστημα μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και ε, Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχω προσωπική άποψη ότι αυτό σπανίως θα αποτελέσει λύση. Θα θέλω λοιπόν εγώ να σας ρωτήσω πώς τοποθετήσετε σε ένα τέτοιο συνδυασμένο συγκεκριμένο σύστημα λύσης και επίσης αντιλαμβάνομαι ότι ε, θα πρέπει να ζητήσουμε ή να προτείνουμε προγράμματα ε, για το μέλλον ε, τι ευρωπαϊκά προγράμματα κατά τη γνώμη σας είναι βασικά και υπάρχουν κατάλληλες δυνατότητες χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επαρκούν οι πόροι για να μπορέσει κανείς να υλοποιήσει τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Θέλετε πρώτα να ακούσουμε μαζεμένες κάποιες ερωτήσεις και μετά να απαντήσετε θέλετε να απαντάτε σε κάθε ερώτηση ξεχωριστά. Γιατί χρόνο έχουμε, αν θέλετε, την κάθε μία χωριστά. Καλύτερα ξεχωριστά την κάθε ερώτηση για να απαντήσω συγκεκριμένα και πιο άμεσα σε κάθε ομιλητή. Σε ό,τι αφορά τη μεικτή συνδυασμένη προσέγγιση Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη στήριξη. Φρονώ ότι η κρίση αυτή είναι η κρίση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν απειλείται η Ελλάδα μόνο, αλλά ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ένωση θα πρέπει να αυτοπροστατευτεί, να υπερασπίσει τον εαυτό της και να δράσει, γιατί είναι δική της η δράση. Είναι πολύ εσφαλμένο να λένε τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης ότι το πρόβλημα είναι ελληνικό, είναι δική τους ευθύνη και αυτοί να πληρώσουν. Αυτό είναι παράλογο για πολλούς και διάφορους λόγους, γιατί ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού χρέους βρίσκεται εκτός της Ελλάδας, σε αλλοδαπά χέρια και αν υπάρξει χρεοστάσιο πάυση πληρωμών, ε, οι ζημίες θα είναι τεράστιες και στη Γαλλία και στη Γερμανία και ίσως ε, μια τέτοια πάυση πληρωμών από μέρου της Ελλάδας απειλήσει τη σταθερότητα πολλών τραπεζών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οποιαδήποτε λοιπόν προσέγγιση που αρνείται το γεγονός ε, ότι η κρίση είναι της Ένωσης και όχι εθνική κρίση της Ελλάδας, ε, κατά τη γνώμη μου οποιαδήποτε προσέγγιση που αρνείται τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα τη κρίση είναι σφαλμένη. Και αν ε, αφήσουν επέμβαση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αντί για την Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήταν λάθος, κολοσιαίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να αποκλειστεί τελείω το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Να χρησιμοποιηθεί και αυτό, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τον κατάλληλο τρόπο. Γιατί η ουσία της διαχείρισης αυτής της κρίσης είναι μια πολιτική διαδικασία και όχι μια τεχνική διαδικασία. Και η πολιτική διαδικασία διαχείρισης της κρίσης, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να γίνει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην ε, επαφεθεί σε ξένα χέρια εκτός της Ένωσης. Ακόμη και αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εγκρίνει κάποιες προϋποθέσεις και όρους που οι περισσότεροι της Ένωσης θεωρούν ανεπαρκείς, δεν θα πιστούν οι αγορές. Οπότε η φήμη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου θα τρωθεί και ούτε η Ελλάδα θα σωθεί. Οπότε σε τελικό βαθμό και σε τελική ανάλυση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αυτή που θα πρέπει κατά κύριο λόγο να διαχειριστεί την κρίση πολιτικά. Και μάλιστα όλα αυτά ήδη περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ε, προηγούμενης διάσκεψης κορυφής της 11ης Μαρτίου. Το κείμενο είναι πολύ σωστά αυτήν την άποψη, πλήρες και προσδιορίζει τις ε, δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς αμφισημίες. Φαίνεται να λένε πολλά αυτά τα συμπεράσματα, αλλά πολύ σωστά αναφέρεται η πρόταση αυτή και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Τώρα, τι, ε, να τι προτίθεται μπορεί να προτείνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλά είναι τα στοιχεία. Μία πρόταση που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φέρει τους G20 στους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς του Bretton Woods. Το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο έχει μια Υπουργική Επιτροπή που είναι το πολιτικό σώμα και μάλιστα υπήρξε και πρόεδρος της πολιτικής αυτής της επιτροπής, της Υπουργικής Επιτροπής όταν ήμουν μέλος της κυβέρνησης. Και είναι, έχει περίπου την ίδια σύνθεση αυτή η Επιτροπή με το G20. Είναι περίπου ίδιες χώρες, οπότε δεν έχει νόημα να υπάρχει το G20 στο οποίο δεν έχει καμία ευθύνη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και οι ίδιοι να συνεδριάζουν στην Διεθνή Επιτροπή Επιτήρησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οπότε οι συζητήσεις που είναι χαρακτηριστικές για το G20 δεν λαμβάνουν χώρα. Οπότε θα μπορούσε να θετηθεί μια τέτοια προσέγγιση ω προ το χώρο συζήτηση. Επίση, θα μπορούσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση να προωθήσει μια συζήτηση για μια καλύτερη δημοσιονομική τάξη. Γιατί αν το δολάριο αποδυναμωθεί, το ευρώ κυρίως θα υποστεί τον κίνδυνο της αναβάθμισης του, της ενίσχυσής του. Κάτι που θα επηρεάσει σοβαρά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων. Οπότε το ευρώ δεν έχει κανένα συμφέρον να υποκαταστήσει το δολάριο. Το αντίθετο, το συμφέρον του ευρώ είναι να δημιουργηθεί μία τάξη παγκόσμια στην οποία κανένα εθνικό νόμισμα και αποκαλώ και το ευρώ εθνικό νόμισμα να είναι η υπερισχύων. Να είναι όλα τα εθνικά νομίσματα τμήματα μιας ε, παγκόσμιας τάξης στην οποία θα ισχύει κοινή διαχείριση. Τέτοιου είδου προτάσεις μπορεί να υποβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπνευσμένη από το δικό της μοντέλο. Και υπερβάμως. Euh, σας ευχαριστούμε κύριε Σόπα. Ήταν πολύ διαφωτιστική και λαμπρή η παρουσίαση σας. Έχω τρεις ερωτήσεις για τη διακυβέρνηση. Μας είπατε προτιμάτε τα φόρα από τους θεσμούς. Τι γνώμη έχετε για το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή την Επιτροπή Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Υπήρξε πρόοδο εκεί. Μήπως θα ήταν ε, σκοπιμότερο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να έχουμε μία δομή που θα αξιοποιεί την εντολή τη σταθερότητας του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Σε ό,τι αφορά την ε, λογιστική εξομάλυνση, πώς θα μπορούσαμε να, τροπη, να τροποποιήσουμε τη διακυβέρνηση, γιατί εκεί έχουμε ένα θεσμό. Αλλά θεσμό αυτορύθμισης. Δεν είναι ούτε φόρουμ, ούτε κανονικός θεσμός, όσο το θέλαμε. Είχαμε προτείνει η ΕΣΒΕ να υπόκειται στο, στην εντολή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου της Παγκόσμιας Τράπεζας ή θα μπορούσαμε να έχουμε και τρίτη οργάνωση. Αλλά το, υπάρχει και το θέμα της ε, λογιστικής εξομάλυνσης που θα πρέπει να εξεταστεί στα πλαίσια της παγκόσμιας διακυβέρνησης. Είπα ότι πιστεύω ότι υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης ε, της διεθνούς νομισματικής τάξης. Τι προτείνετε για να σημειωθεί πρόοδος εκεί. Γιατί όταν οι δύο Ζαν Κλοντ και ο Επίτροπος πάει στην Κίνα, είναι σαν να, μεταφέρει, είναι, σαν να είναι αγγελιοφόροι των Αμερικανών. Πώς θα μπορούσε και η Ευρώπη να υψώσει τη φωνή της εκεί και να μην γίνει το μπαλάκι του πινκ-πονγκ μεταξύ Αμερικανών και Κινέζων. Από άποψη παγκόσμια δικυβέρνηση αυτό το θέμα μας απασχολεί ιδιαίτερα. η Επιτροπή, το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η Επιτροπή άλλαξε το όνομα, αλλά όχι η λειτουργία. Επεκτάθηκε και στο G20, δηλαδή παρακολούθησε αυτή τη μετάβαση από το G7 ή G8 στο G20 ως προς τη σύνδεση, αλλά παρέμεινε φόρουμ. Δηλαδή, δεν συνοδεύεται από μια νομική βάση, δεν έχει δική του δομή, ούτε έχει κύρος εφάμιλο με του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου ή της Παγκόσμιας Τράπεζας. Έχει και γραμματεία, που είναι λίγο μελής σε σχέση με το καθήκον που έχει να επιτελέσει και σε σχέση με τη γραμματεία του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου της Κεντρικής Τράπεζας. Πάντως είναι χρήσιμο αυτό το όργανο γιατί μόνο εκεί, μόνο στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ή στο Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας μπορούν να μιλήσουν διάφοροι φορείς, κεντρικές τράπεζες, ε, ε, οργανισμοί επιτήρησης, υπουργοί Οικονομικών που δεν είχαν την ευκαιρία να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι. Πάντως καλό θα ήταν ο οργανισμός αυτός να προσαρτηθεί με πιο πάγιο τρόπο στους θεσμούς που ανέφερα προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο μπορεί να κάνει το ίδιο έργο με το φόρουμ της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας. Και υπάρχει ένας καταμερισμός των ρόλων πολύ πιο σαφής τώρα. Το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο είναι αρμόδιο για να τηρηθούν επιτόπου οι κανόνες. Σε ό,τι αφορά τις, τους λογιστικούς κανόνες, γνωρίζω τις ευρωπαϊκές επιφυλάξεις ως προς το ΙΑΣΚ, και εγώ αναμίχθηκα ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, το ΙΑΣΚ. Πιστεύω ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να είναι υπερήφανοι για το ΙΑΣΚ αντί να παραπονιούνται. Και οι... αυτοί που θέτουν τι προδιαγραφέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι οι ίδιοι που το κάνουν και διεθνώ. Και αν αυτό συνέβαινε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ε, θα υψωνόταν εδώ κατακραυγή κατά του Αμερικανικού Ιμπεριαλισμού. Το, αυτό κάνουμε εμεί, αλλά παραπονιόμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Δεν είναι αλήθεια ότι επιβάλλονται κάποιοι κανόνες από τους ε, διαμορφωτές των προδιαγραφών χωρίς ευθύνες και χωρίς ε, λογοδοσία. Οι κανόνες ISB δεν ε, αποκτούν δεσμευτικό χαρακτήρα αν δεν δοθεί το πράσινο φως από τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και η διαδικασία επιστοποίησης είναι ε, η ίδια διαδικασία που ισχύει για την μεταμόρφωση μιας πρότασης σε κανονισμό. Κάτι αντίστοιχο ισχύει στις Ηνωμένες Πολιτείες με το FASB. Το αντίστοιχο όμως ευρωπαϊκό όργανο είναι και ο παγκόσμιος της προδιαγραφών. Πολύ περισσότερο από το FASB των Ηνωμένων Πολιτειών. Βέβαια θα μπορούσαν να γίνουν κάποιες βελτιώσεις, αλλά το να το θεωρήσουμε ως ανομαλία που θα πρέπει να καταργηθεί δεν είναι σωστό. Είναι βέβαια κάπως περίεργο ώστε να είναι μόνο Ευρωπαίοι αυτοί που καθορίζουν ε, τις προδιαγραφές και τους κανόνες. Αλλά άμα θέλει κανείς έχει πρωταγωνιστικό ρόλο και να λύνει και να δένει διεθνώς, ε, θα πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Σε ό,τι αφορά την παγκόσμια ε, νομισματική τάξη, δεν μπορώ να σας απαντήσω μέσα σε μισό λεπτό. Πάντως και μόνο που διαπιστώνουμε ή αποδεχόμαστε το συμπέρασμα ότι στο μέτρο που το παγκόσμιο νόμισμα είναι εθνικό νόμισμα, υπάρχει μία θεμελιώδης αντίφαση μεταξύ της ανάγκης της νομισματικής πολιτικής του, της χώρας που έχει αυτό το νόμισμα και των το, νομισματικών αναγκών του υπόλοιπου κόσμου. Και μόνο αυτή η αποδοχή του, αυτού του συμπεράσματος είναι αρκετό αρκετή. Δεν θα υπάρξει παγκόσμια νομισματική τάξη υποφερτή αν δεν υπάρξει νέο νόμισμα. Κάτι που είχε για 40 χρόνια που τέτοιο ρόλο έπαιζε ο Χρυσό. Δεν προτείνω βέβαια επαναφορά του χρυσού, αλλά υπήρχε ένα παγκόσμιο γνώμονα μέχρι το 1971 και ήταν ε, ο Χρυσό. Ο, Ρι... ο Ρομπέρτ Τριφέν πριν από 50 χρόνια κατέδειξε αυτή την αντίφαση. Και η σημερινή κρίση, για πολλούς και διάφορους λόγους, είναι η συνέπεια αυτής της α, ε, θεμελιώδους αντίφασης. Και τώρα, αν με ρωτάτε πώς θα ξεφύγουμε από αυτή την αντίφαση, την ίδια ερώτηση μου είχε κάνει και ένας δημοσιογράφος και το απάντησα εγώ μπορώ να σας κάνω την επίδειξη ότι χρειαζόμαστε ένα αντικείμενο που να πετάει, αλλά δεν έχω, δεν έχω εφεύρει ακόμη το αεροπλάνο. Το γεγονός όμως ότι δεν έχουμε ακόμη το αεροπλάνο δεν σημαίνει ότι η επίδειξη ή η η πρόταση ότι χρειαζόμαστε ένα υπτάμενο αντικείμενο είναι σφαλμένη. Υπάρχουν κάποια πιθανά όργανα, να, δούμε και ένα σύστημα συναλλαγών. Πάντως, στον τομέα αυτό θα πρέπει να βρούμε τις λύσεις. Αλλά να συμφωνήσουμε καταρχήν ότι χρειαζόμαστε λύση, ότι χρειαζόμαστε αυτό το υπτάμενο αντικείμενο. από τις Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου μοιάζει με αυτή της κυρίας Περές. Υπάρχει τεράστια ανισορροπία, όπως είπατε κι εσείς. Και επισημάνατε την έλλειψη περιορισμών για τις ΗΠΑ. Δεν ισχύουν οι ίδιοι περιορισμοί με τους, για τους Αμερικανούς με εμά, γιατί εμείς έχουμε μηχανισμούς που μας επιτρέπουν να επανέλθουμε στο σωστό δρόμο όταν διαπιστώνουμε ανισορροπίες. Είπατε ότι η Ευρώπη θα πρέπει να εξαγάγει το μοντέλο της για να τερματιστεί αυτή η αλλοπρόσαλη κατάσταση. Αυτό το καταφέραμε στην Ευρώπη. Δηλαδή καταργήθηκαν χάρη στο ενιαίο νόμισμα οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις νομισμάτων, αλλά γι' αυτό χρειάστηκε να καταρρεύσει ολόκληρο το τείχος του Βερολίνου. Και αν χρειαζόταν να ξανακάνουμε κάτι τέτοιο το 2010, με τέτοια μετριοπαθή πολιτική βούληση. Πολύ φοβάμαι ότι δύσκολο θα ήταν ε, σήμερα να υλοποιήσουμε την παλιά υπόσχεση. Επίσης είπατε ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρωτοστατήσει στη συζήτηση για την αναθεώρηση της, ε, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, για τη μεταρρύθμιση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η θεωρία σας για τα φόρα είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Υπάρχουν όμως και άλλα φόρα, ο για παράδειγμα, Μήπως θα μπορούσαμε τη ζήτηση αυτή να τη μεταφέρουμε και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Πιστεύετε ότι για να σταματήσουν αυτές οι ανταγωνιστικές υποτιμήσεις ή χρόνιες υποτιμήσεις του δολαρίου για παράδειγμα και του κινέζικου νομίσματος. Δεν πιστεύετε ότι... Γιατί για το εμπορικό dumping ε, να πούμε ότι δεν είναι, δεν είναι αποδεκτό στον ΠΟΕ κάτι τέτοιο να ισχύσει για τα χρόνια υποτιμημένα νομίσματα. Δηλαδή να μεταφέρουμε αυτή τη συζήτηση και στην Παγκόσμια Οργάνωση Εμπορίου. Ερωτώ λοιπόν, πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μπλοκάρει τις διαπραγματεύσεις Ντόχα έως ότου βρεθεί λύση για την κατάσταση αυτή. Να προσθέσω πως είχα θέσει ακριβώς την ίδια ερώτηση στον κύριο Τουπουασέ πριν από ένα χρόνο περίπου και μου είπε ότι αν μπείτε σε ένα φόρουμ και χτυπήσετε τους Κινέζους η διάσκεψη τελειώνει μέσα σε 10 λεπτά. Εγώ δεν είμαι υπέρ του μπλοκαρίσματος. Η διαδικασία της Ντόχα, κατά την άποψή μου, θα πρέπει να συνεχιστεί και θα πρέπει να προσθεθούν πράγματα και όχι να αφαιρεθούν μέσα στη διαδικασία προσπάθειας διαχείρισης της διεθνούς ολοκλήρωσης. Είναι αλήθεια ότι δεν υπάρχει κάποιος χώρος όπου να μπορούμε να συζητήσουμε πλήρως τις σχέσεις των, ε, των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τη σχέση αυτών με τις εμπορικές ε, σχέσεις. Τα τρία όργανα τα οποία είχαν φτιαχτεί στη δεκαετία του 40, ο ΠΟΕ έγινε πολύ αργότερα γιατί ε, η χάρτα της ε, Βάνας, την οποία είχαμε διαπραγματευτεί το δεκαετία του 40, δεν επικυρώθηκε από το Αμερικανικό Κογκρέσο και άρα το μεταπολεμικό σύστημα δημιουργήθηκε χωρίς έναν από τους τρεις προβλεπόμενους πυλώνες. Η Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο που είναι και τα τρία μέσα στο ε, πλαίσιο ε, του ΟΗΕ θα έπρεπε να συνδεθούν σε ένα επίπεδο ώστε να μπορούμε να συζητήσουμε και να αναζητήσουμε συμφωνίες που να ε, περνούν από τον ένα τομέα στον άλλον, όπως συνήθως γίνεται δηλαδή ανάμεσα στο νόμισμα, στις ισοτιμίες και στο εμπόριο. Σήμερα κάτι τέτοιο δεν γίνεται. Ναι, συμφωνώ ότι μπορούμε να κάνουμε τέτοιου είδου συζήτηση και στον ΠΟΕ. Θα πρέπει ωστόσο να αναπτυχθεί περισσότερο και στον Δούνο και από τη στιγμή που υπάρχει μια συζήτηση ανάμεσα στους ε, ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων, όλα αυτά τα θέματα θα συζητιώνται γιατί συνδέονται μεταξύ τους. Κυρία να σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ για αυτήν την ε, πολύ ενδιαφέρουσα εισήγηση. Η ε, και εγώ σκεφτόμαστε, ε, μου φαίνεται με τον ίδιο τρόπο, γιατί οι τρεις ερωτήσεις που είχα εγώ καταγράψει ήδη τέσσερα από την υπερβάνωση, διαβάζουμε τα ίδια βιβλία, δεν ξέρω, τα ίδια κείμενα. Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να αναφερθώ σε κάτι που είπατε, ότι δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως ένα πρότυπο για την παγκόσμια διακυβέρνηση σε σχέση με τα θεσμικά όργανα και ίσως ε, να δούμε πώς θα φάλουμε τάξη στα του οίκου μας καταρχήν, γιατί συμφωνώ ότι οι θεσμοί και όχι τα φόρα είναι περισσότερο ο τρόπος για να προχωρήσουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, αλλά έχω την αίσθηση πως το ευρωπαϊκό πρότυπο διακυβέρνηση δεν ήταν το καλύτερο δυνατό κατά τα τελευταία χρόνια. Και σίγουρα έχουμε κάποια κριτήρια τα οποία περιγράφει το Μάστριχτ και τα περισσότερα κρατημέλη έχουν ε, παραβιάσει αυτά τα στάνταρ. Και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα μάλιστα. Φαντάζομαι πως το θέμα είναι λοιπόν πώς θα αλλάξει η νοοτροπία των κρατών μελών. Η νοοτροπία συμμόρφωσης προς κανόνες τους οποίους ήδη έχουν συμφωνήσει. I I am very strongly convinced that the process of uh, keeping one owns house in order. Πιστεύω όντως πως το να βάλουμε τάξη στα του οίκου μας ή να επιβάλλουμε τους ισχύοντες κανόνες στις χώρες μας δεν θα πρέπει να θεωρηθεί ως προϋπόθεση για να αρχίσουμε να λειτουργούμε και να συνεργαζόμαστε με άλλες χώρες. Όχι. Το να έχουμε αυτή την ιδέα όπως είναι αυτό προϋπόθεση είναι πολύ επικίνδυνο κατά την άποψή μου τόσο εντός περιφερειακών ενώσεων όπως η Ένωσή μας, όσο και στο πλαίσιο του παγκόσμιου συστήματος. Ποτέ κανένα σπίτι δεν, είναι, δεν βρίσκεται σε απόλυτη τάξη. Και η τάξη πάντοτε μπορεί να διαταραχτεί από την ταξί που επικρατεί στο διπλανό σπίτι και είναι πολύ δύσκολο να πει κανεί πού αυτό ξεκινά και πού τελειώνει. Η Ένωση δεν έχει εξωτερικές, ε, σημαντικές εξωτερικές ανισορροπίες. Είμαστε βέβαιοι πως αν οι εξωτερικές ενισορροπίες των ΙΠΑ και του να διορθωθούν θα παραμείνει η Ένωση χωρίς ανισορροπίες ή μίσως στο πλαίσιο της περιφερειακής και παγκόσμιας προσαρμογής θα βρεθεί η Ένωση με προβλήματα. Δεν το ξέρουμε, γιατί είναι τόσο περίπλοκα τα πράγματα που δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τέτοιο δεχόμενο. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εξωτερική ανισορροπία, αλλά έχει τεράστιες εσωτερικές ε, ανισότητες, όπως είδαμε σήμερα. Εάν θεωρούμε πως η τάξη σημαίνει πλεόνασμα, είναι αδύνατον όλοι να έχουν πλεόνασμα. Κανένας δεν θα έλεγε πως ένα πλεόνασμα είναι ένδειξη αταξίας, αλλά αν το έλλειμμα είναι ένδειξη αταξίας θα πρέπει να δεχτούμε ότι εάν διορθώσουμε την αταξία θα πρέπει να διορθώσουμε ε, και ε, αυτούς που έχουν πλεόνασμα. Χρειάζεται δηλαδή να υπάρξει κάποια αλληλεπίδραση. Εγώ πιστεύω και είπα ότι ε, αν η Ένωση έπρεπε να εφαρμόσει καλύτερα το μοντέλο της, θα είχε πολύ περισσότερο κύρος ώστε να το προτάξει ως ένα συνδυασμό κάποιων βασικών αρχών που είναι κατάλληλοι για παγκόσμια διακυβέρνηση. Γιατί είναι αρχές για τη διαχείριση της αλληλεξάρτησης. Και αυτό είναι και το κλειδί, η αλληλεξάρτηση. Εάν όμως περιμένουμε πρώτα να τα τακτοποιήσουμε όλα, δεν θα κινηθούμε ποτέ. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο να κάνουμε ακόμη ένα γύρο ερωτήσεων. Επανέρχομαι στο ΕΛΚ. Ποιος θα ήθελα να κάνει κάποια ερώτηση. Σας ευχαριστώ. Αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι γιατί δεν θεωρούμε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ως ένα θεσμό που μπορεί να βοηθήσει οποιαδήποτε χώρα, είτε αυτή ανήκει στην Ευρωζώνη είτε όχι. ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με κάποιες χώρες της Ένωσης ήταν πολύ καλός, δηλαδή ταχύς, συγκεκριμένος, ακριβής και έδωσε και αποτελέσματα. Και δεν καταλαβαίνω γι' αυτό γιατί δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν θεσμό που είναι ε, ειδικευμένος στην αντιμετώπιση προβλημάτων ε, χωρών με τέτοια με ελλείμματα. Γιατί δεν αφήνουμε λοιπόν το Διεθνέ Μησοδοτικό Ταμείο να κάνει τη δουλειά του. Δεν ξέρω αν μιλάτε για μένα ή για, σε μένα ή απευθύνεστε σε μένα ή σε κάποιον άλλον. Εγώ πιστεύω πως ε, υπάρχουν δύο θέσεις οι οποίες ε, κατά την άποψή μου είναι λανθασμένες. Η μία είναι ότι ο ΠΟΕ ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να παίξουν, να αποκλειστούν τελείως από οποιαδήποτε πτυχή χειρισμού ή διαχείριση της ελληνικής κρίσης. Και η άλλη επίση λανθασμένη θέση είναι ότι το πρόβλημα τη ελληνική κρίση είναι κάτι το οποίο μπορεί να αγνοήσει τελείω η Ένωση, δεν την αφορά. Θα πρέπει να απασχολήσει μόνο το Δουνουτού, όπω θα απασχολούσε και οποιαδήποτε άλλη από τι κόσμο. Και οι δύο αυτέ ε, θέσει είναι λανθασμένε κατά την άποψή μου, γιατί η Ένωση είναι κάπου στο μέση. Δηλαδή δεν είναι ακριβώ όπω είπα. Αλλά η Ελλάδα είναι για την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει για την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πολύ περισσότερο από ό,τι οποιαδήποτε άλλη χώρα εκτός ε, της Ευρωζώνης. Αν το, η πολιτεία της Καλιφόρνιας που έχει πολύ σοβαρά προβλήματα δημοσιονομικά. Εάν ε, ε, αντιμετώπιζε κίνδυνο κρίσης, τότε η Ουάσιγκτον, το Κογκρέσο, και η Αμερικανική κυβέρνηση θα αντιμετώπισαν και θα βοηθούσαν τον πολιτεία. Και όλοι θα θεωρούσαν πω ε, ήταν αυτό απόλυτα φυσιολογικό. Κανένα δεν θα στρεφόταν στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο. Η Ελλάδα δεν είναι η Καλιφόρνια, ευτυχώ. Ε, γιατί είναι αυτό πολύ πιο καλό για την Ένωση. Αλλά όπως σας είπα, η Ένωση είναι Ένωση. Δεν είναι απόλυτη Ένωση, δεν είναι πλήρως ενωμένη, αλλά έχει ενιαίο νόμισμα, έχει ολοκληρωμένο χρηματοπιστωτικό σύστημα και επειδή το ελληνικό χρέος είναι στα χαρτοφυλάκια πολλών τραπεζών εκτός Ελλάδος, δηλαδή οι αποταμιεύσεις πολλών Γερμανών, Γάλλων και Ολλανδών είναι επενδεδημένες σε ελληνικούς τίτλους, το να θεωρήσουμε ότι ο χειρισμός της ελληνικής κρίσης σημαίνει πως κάνουμε χάρη στην Ελλάδα, όχι, καθόλου δεν πρόκειται περί αυτό. Το να βοηθηθεί μια χώρα να βγει από την κρίση ώστε να διασφαλιστούν οι πιστώσεις με τα κατάλληλα μέτρα δεν βοηθά μονάχα την Ελλάδα, βοηθά ολόκληρη την Ένωση. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν νομίζω πως η Ένωση δεν μπορεί να μείνει εκτός αυτό που είναι υποαπειλή είναι η, ενο... η ενότης της Ένωσης. Αν λοιπόν αυτό γίνει αποδεκτό, ε, τότε το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο μπορεί να παίξει ρόλο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Ένωση. Κύριος Μπονσινιόρε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Μια ερώτηση, Πρόεδρε. ποιο μέσο θα βλέπατε για να δώσετε συνέχεια στη δική σας ε, σκέψη παρέμβαση της Ένωσης. Πιστεύετε πως θα ήταν πιο χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό νομισματικό ταμείο ή θεωρείτε πιο σωστό, όπως λένε ορισμένοι, ότι δεδομένου ότι πρέπει να παρέμβει κανείς και σε διμερές επίπεδο για να λυθεί το πρόβλημα. Ευχαριστώ. ένα Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και θα χρειάζονταν χρόνια για να δημιουργηθεί κάτι τέτοιο. Ίσως λοιπόν να ήταν καλή ιδέα να δημιουργηθεί, αλλά για την ώρα, για την ελληνική κρίση δεν εξυπηρετεί τίποτα. Αυτό δεν σημαίνει πως ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί συλλογικά να δημιουργήσει ένα είδος συλλογικής στήριξης. Αυτή τη στιγμή η εναλλακτική είναι ανάμεσα στην ε, συλλογική στήριξη της Ένωσης και τη στήριξη από κάποιες χώρες. Σίγουρα θα ήταν καλύτερο να υπάρξει μια συλλογική στήριξη από πλευρά της Ένωσης. Όμως δεν νομίζω πως από αυτού θα πρέπει να είμαστε εξαιρετικά άκαμπτοι. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι οι συνθήκες εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας, τα κίνητρα, η πολιτική στήριξη προς αυτές τη, αυτή την δράση εξυγένσης να προέλθουν από την Ένωση. Αν στη συνέχεια μέσα σε αυτό το πλαίσιο διάφορα μέτρα ληφθούν από κάποιες χώρες αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο διαχείρισης της κρίσης από πλευράς της Ένωσης ή αν προερχόταν αυτή η, από όλε τι χώρε, κατά την άποψή μου δεν έκανε μεγάλη διαφορά. Επανέρχομαι στους σοσιαλιστές. Δεν ξέρω αν η, η κυρία Γιακονσάβη θέλει να κάνει μία ερώτηση. Ευχαριστώ. όσον αφορά την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση και την ε, ε, επί τις επιπτώσεις της κρίσης στην αναπτυσσόμενες χώρες. Μπορείτε να μας πείτε ποια θα είναι η αντίκτυπος της κρίσης στην Κένια ή οποιαδήποτε άλλη χώρα, αν θέλετε. Κοιτάξτε, μην νομίζετε ότι είμαι τόσο εμπειρογνώμονας. Δεν ξέρω. Μα εν γέννη μπορείτε εσεί να αναπτύξετε τι είδους αντίκτυπο θα έχει αυτή η κρίση στι αναπτυσσόμενες χώρες. Κοιτάξτε, υπάρχουν τρεις ομάδες χωρών. Οι προηγμένες οικονομίες, οι, αν, οι οικονομίες και οι χώρες χαμηλού εισοδήματος στον κόσμο. Για τις προηγμένες οικονομίες, βασικά Ευρώπη, είπα η Ιαπωνία, ίσως και κάποιες ακόμα Κορέα και μια-δυο ακόμα, κατά την άποψή μου η κρίση θα οδηγήσει σε σημαντική μείωση του ποσοστού μεγέθυνσης της οικονομίας για τα επόμενα χρόνια. Για τις αναδυόμενες οικονομίες δεν νομίζω πως η μεγέθυνση θα περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό και το βλέπουμε ήδη αυτό. Βραζιλία, Κίνα, Ινδία. Μεγεθύνει την οικονομία τους ε, σε ποσοστά πάνω του 5% και πολλέ φορέ φτάνουν και στο 10%. Και αυτό γιατί η μεγέθυνση εκεί ε, βασίζεται στο να βγουν από τη φτώχεια. Δηλαδή, εκείνοι δεν έχουν ακόμα πράγματα τα οποία να πετάνε. Εμείς αντικαθιστούμε αυτοκίνητα, τηλεοράσεις και ούτω καθεξής, ενώ ακόμα λειτουργούν. Στην Κίνα βρίσκονται στο στάδιο του να αγοράσουν για πρώτη φορά αυτοκίνητο ή, ή σπίτι. Αυτό είναι μια διαδικασία κοινωνική αλλαγή που δεν θα σταματήσει κατά την άποψή μου λόγω τη κρίση. Και έπειτα υπάρχουν και οι χώρε χαμηλού εισοδήματο Ορισμένες από αυτές μπορεί και να μετακινηθούν στο στρατόπεδο των αναδειωμένων και εκεί είναι πιο δύσκολο να προβλέψει κανείς. Και πάλι αυτές οι χώρες χτυπήθηκαν λιγότερο γιατί δεν είχαν και τίποτα για να χτυπηθεί. Αλλά εν αν καιρό αυτή η κρίση προκάλεσε σημαντική, αν μάλλον αυτή η κρίση οδηγήσει σε σημαντική επιστροφή στο προστατευτισμό, θα ήταν καταστροφικό για αυτές τις χώρες σε σχέση με το θέμα, ας πούμε αυτό που αναφέρθηκε πριν για μπλοκάρισμα του γύρου της Δόχα. Αν ολοκληρωθεί επιτυχώς ο γύρος της Δόχα, ορισμένε από αυτές τις πολύ φτωχές χώρες θα μπορούσαν να εξάγουν ε, προϊόντα κλωστηφαντουργίας, να αρχίσουν μια διαδικασία δηλαδή που να τους βοηθήσει. Δεν γνωρίζω ακριβώς ε, λοιπόν τι θα συμβεί με αυτές τις χώρες, αλλά για την ώρα να σας πω ότι δεν ήταν αυτές που χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση. Μπορεί όμως να χτυπηθούν σε μια δεύτερη φάση. Uh, εγώ θα ήθελα να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις. Ω τελευταίο βουλευτή εδώ σε αυτό το γύρο, εγώ θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η δική σα αξιολόγηση της προσέγγισης για το G20 ξεκίνησε πριν από 1,5 χρόνο και είχαμε όλοι πολύ μεγάλες προσδοκίες. Εγώ προσωπικά έχω απογοητευτεί από το τι έχει συμβεί μέχρι στιγμή και έχω εγκαταλείψει την ελπίδα πως πραγματικά θα δώσουν μια παγκόσμια απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις που προέρχονται από την κρίση. Θα υπάρξει μια απάντηση από την Ευρώπη, μια απάντηση από την Αμερική και ούτω καθεξής. Δεύτερο σημείο. Η κρίση νομίζω ε, δίδαξε στους Ευρωπαίους πως εκτός του ότι υπάρχει ένα ενιαίο νόμισμα ότι είμαστε δηλαδή μια νομισματική ένωση, θα πρέπει να καταφέρουμε να έχουμε πολύ στενότερη συνεργασία στην οικονομική πολιτική, στη φορολογική πολιτική και ίσως και να πρέπει να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. νομίζω όμως ότι όλα αυτά δεν έχουν καταστεί απόλυτα σαφή για τον κόσμο. Και έπειτα, για να μπορούμε να βγούμε από τέτοιε δύσκολε καταστάσει όπω το τεράστιο δημόσιο έλλειμμα, χρειάζεται μεγέθυνση. Ανάπτυξη και ανάπτυξη που να είναι τουλάχιστον τόσο ψηλή όσο αυτή που κρίνουμε ότι είναι η δυνητική μα ε, ανάπτυξη. Ερώτησή μου λοιπόν είναι, βλέπετε να υπάρχει ο πειρασμός από τη στιγμή που δεν μπορούμε να καταφέρουμε την ανάπτυξη ανάπτυξη αυτή να προσπαθήσουμε να λύσουμε το πρόβλημα μέσω του πληθωρισμού. Μου δίνετε μια ώρα για να απαντήσω. Για την πρώτη σας ερώτηση. Όπως είπα, νομίζω πως το G20 ήταν ένα βήμα μπροστά σε σχέση με το G7. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να συγχωνευτούν αυτά που εγώ αποκαλώ φόρα σε θεσμούς. Αλλά και αυτό δεν θα αρκέσει. Το ερώτημα που θέσατε, που νομίζω ότι είναι αρκετά κέριο, είναι οι μεταρρυθμίσεις τελικά θα συμφωνηθούν διεθνώς ή σε εθνικό επίπεδο ή θα είναι τοπικές μεταρρυθμίσεις. Νομίζω πως είναι ακόμα ανοιχτό το τι θα γίνει. Ίσως στο τέλος ε, οι μεταρρυθμίσεις να είναι βασικά εθνικές και τοπικές και ίσως να υπάρχει ακόμα λιγότερη ομοιομορφία κανόνων στην παγκόσμια οικονομία από ό,τι σήμερα. Για παράδειγμα, η η χρηματοπιστωτική μεταρρύθμιση συζητάται συζητάτε στο φόρουμ για την ε, δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά μετά ο καθένας βγαίνει και κάνει τις δικές του ανακοινώσεις. Ακόμα και η Ένωση βρίσκεται σε φρικτή κατάσταση και μπορώ να σας το πω γιατί το γνωρίζω άμεσα πως ξέρετε τι είναι το ΣΕΜΣ. ΣΕΜΣ. Το, στο ΣΕΜΣ γίνονται συνεδριάσεις όπου η ευρωπαϊκή α, θέση συντονίζεται εν ώψη του G10. Κάθε ευρωπαϊκή χώρα λέει τις απόψεις της εκεί και ξεχνά τελείως ποια είναι η κοινή θέση που αποφασίστηκε στο ΣΕΠΣ. Αυτή είναι μια ε, περίπτωση λοιπόν όπου η Ένωση δίνει το κακό παράδειγμα και όχι το καλό. Ο κίνδυνος λοιπόν μεγαλύτερου κατακαιρματισμού αντί για περισσότερη ομοιομορφία ή συνοχή στους διεθνούς κανόνες νομίζω ότι είναι πολύ ψηλός. Έπειτα και η συνεργασία της μεγαλύτερη σε άλλους τομείς, εκτός δηλαδή από την νομισματική πολιτική. Στον ε, νομισματική πολιτική, αυτό που έχουμε στην Ευρώπη δεν είναι συνεργασία, είναι ένωση. ενώτης. δηλαδή συνεδριάζουν στην Φραγκφούρτη και, και προκύπτει μια απόφαση ακόμα και αν δεν έχουν διαφωνήσει μεταξύ τους. Δεν είναι όπως αυτό που συμβαίνει εδώ συχνά, όπου αν δηλαδή διαφωνούν όλοι πάει ο καθένα σπίτι του και κάνει το δικό του. Ε, αν η νομισματική πολιτική γινόταν με αυτόν τον τρόπο, τότε ο κόσμος θα γελούσε μαζί μας. Εδώ λοιπόν δεν μιλάμε για συνεργασία ή ακόμα και για δομημένη συνεργασία ή για συντονισμό. Είναι ένωση, ενότητα και για να υπάρχει ενότητα θα πρέπει να ενεργούμε με τα ευρωπαϊκά μέσα και όχι απλά να έχουμε την ε, ε, βούληση να συντονίζουμε τα εθνικά μέσα. Αυτά τα κάνουν κυβερνήσεις. Τα ευρωπαϊκά όμως μέσα είναι πολιτική της Ένωσης υπάρχει μια ε, βούληση για συνέχιση, για συνέχεια. Αν δούμε πώς λειτουργούν τα ομοσπονδιακά κράτη, ομοσπονδία δεν παρεμβαίνει στα κράτη. Εδώ δεν θέλουμε ομοσπονδία, αλλά θέλουμε να παρέμβουμε. Νομίζω πως αυτό είναι λάθος. λιγότερο θα πρέπει να προσπαθούμε να συντονίσουμε τα κράτη-μέλη και να έχουμε μεγαλύτερη διάθεση ώστε να ενεργοποιήσουμε τα μέσα τα κοινοτικά σε πολλού τομεί που βρίσκονται στη συνθήκη, δηλαδή έρευνα, περιβάλλον, μεταφορέ, υποδομέ, ενέργεια. Για όλου αυτού του τομεί θα έπρεπε να υπάρχει ένα κομμάτι, γιατί αυτά είναι κοινέ αρμοδιότητε, να είναι ένα κομμάτι όπου η η, η Ένωση να παίζει ρόλο ενεργό, όχι συντονιστικό. Ναι, ίσως κάποια στιγμή να πρέπει να υπάρξει πληθωρισμός για να βγούμε από την κρίση και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η ελληνική κρίση είναι τόσο σημαντική. η μεγαλύτερη, ε, το μεγαλύτερο φρένο για, κατά του πληθωρισμού αυτή τη στιγμή είναι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Γι' αυτό και έχει πιεστεί τόσο η ελληνική κρίση, ώστε τελικά να έχει υποβαθμιστεί η δύναμη του ευρώ και της νομισματικής ένωσης. Και αυτό είναι ένα βήμα προς την πληθυριστική λύση. Γι' αυτό και πιστεύω ότι για τη Γερμανία είναι τόσο σημαντικό παρά τα όσα διαβάζουμε ορισμένες φορές στον τύπο να λάβει υπόψη ότι η ελληνική κρίση αποτελεί απειλή για την σταθερότητα τιμών και στη Γερμανία. Και θα ήταν μια τεράστια χάρη για αυτούς που θέλουν ε, λιγότερο ισχυρή υπεράσπιση της σταθερότητας των τιμών και ισχυρότερη αντίσταση στην πληθωριστική λύση, να πούνε δηλαδή ότι η Ελλάδα πρέπει να αφαιθεί στη μοίρα της. Ευχαριστώ. Έτσι ολοκληρώσαμε αυτό το πρώτο μέρος και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή εν ονόματι όλων σας για, τα, για τις ε, δηλώσεις του διότι ήταν πάντοτε πολύ φωτισμένη η παρουσίασή του και προχωράμε τώρα στο επόμενο θέμα.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 προσέξετε διότι τώρα ερχόμαστε στο δεύτερο μέρος της ε, συνεδριάσεώς μας. Στην αρχή μιλήσαμε για τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Ε, τώρα ε, σε αυτό το θέμα έχουμε τρεις σημαίνουσες προσωπικότητες. Καταρχήν τον κύριο Μπέρτ Βαντσέλμ διότι έχετε όμως τα βιογραφικά τους. Ο κύριος Βαντσέλ είναι από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δίπλα είναι ο Σόνι Καπούρ ενός think tank, μία ομάδας συλλογισμού που λέγεται Redefine και ε, συζητάνε την αναμόρφωση των δημοσιονομικών θεμάτων της διακυβέρνηση κτλ. Και τρίτος ο Στέφαν Σουλμάιστερ από το Αυστριακό Ινστιτούτο Οικονομικής Έρευνας. Ε, θα σας δώσω το λόγο και θα σας παρακαλούσα σε 10 λεπτά ο καθένας από εσά να παρουσιάσει το θέμα του. Σας ευχαριστώ. Είναι μεγάλη χαρά για μένα εδώ και βλέπετε ότι ο τίτλος μου της ομιλίας μου είναι πολύ μακρύς πώς θα διορθώσουμε τον κόσμο στα γρήγορα αλλά εδώ βλέπετε ε, έχω λίγο χρόνο στη διάθεσή μου και γι' αυτό θα σας μιλήσω σύντομα για την κρίση, τι κάναμε και μετά θα βασιστώ στον κόσμο μετά την κρίση. Ε, ε, εάν θα υπάρχει μια αναμόρφωση του G20 του Διεθνούς Νομισματικού Συστήματος και ο προλαλής σας ε, είπε πολλά σοφά πράγματα για αυτά τα θέματα οπότε εγώ θα προσπαθήσω απλώ να συμπληρώσω. Όπως σας είπα η κρίση ήταν τρομερή, συγχρονισμένη, βαθιά, ολοκληρωμένη νομίζω ότι μου λείπει μία διαφάνεια. Κρίμας. Διότι θα σας έδειχνα πόσο κακή είναι η κρίση, αλλά τέλος πάντων. Εδώ το, θα το βρείτε στο έγγραφο που βλέπετε το 2009 είναι ε, εκτός όλων των δυνατοτήτων. Το 2010 φαίνεται κάπως καλύτερα και είναι κάπως βελτιωμένο σε σχέση με το 2009. Ε, εδώ λοιπόν ε, όπως βλέπετε υπάρχουν πολλά οικονομικά στοιχεία υπήρξε χρηματοδότηση 170 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ε, υπήρξαν και άλλες μεταρρυθμίσεις στις οποίες θα αναφερθώ ε, και θα ήθελα να σας πω πού προσγειωνόμαστε ε, και τι γίνεται με την εποπτεία και με τον πολιτικό διάλογο. Ε, τώρα βλέπετε ε, μία συγκέντρωση ε, τον δανεισμό από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο το οποίο συνέβαλε πολύ στην κάλυψη της κρίσεως χώρες οι οποίες διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να έχουν προχωρήσει τα προγράμματα ήταν ευέλικτα όχι μόνο για να καλύψουμε ε, τα ε, ελλείμματα των ισοζυγίων πληρωμών αλλά και των προϋπολογισμών. Τους είπαμε επίσης, τους υποδείξαμε πώς θα χρησιμοποιούσαν αυτά τα χρήματα και τα αποτελέσματα είναι καλά. Δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις όπου εφαρμόσαμε ένα πρόγραμμα είδαμε ότι η οικονομική κατάσταση βελτιώθηκε. Λοιπόν, όχι μόνο αλλάξαμε τα ποσά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο δανείζουμε, εδώ θα ήθελα να τονίσω ότι έχουμε μία ευέλικτη γραμμή πιστώσεως ε, και εδώ πρόκειται για μεγάλη, για μεγάλη δυνατότητα πιστοληπτικής δυνατότητας ε, για ορισμένες χώρες ε, το χρησιμοποιήσαμε στην Κολομβία όπου δεν χρησιμοποίησαν τα χρήματα αυτά αλλά έδωσαν ένα σωστό μήνυμα στην αγορά ότι ε, αν χρειαζόντουσαν η χρηματοδότηση υπήρχε και αυτό είναι κάτι το οποίο θα κάνει και στο μέλλον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Επίσης όπως είπε και ο προλαλής σας, εμείς δανείσαμε 280 δισεκατομμύρια εκατομμύρια δολάρια. Δεν θα προσπαθήσω τώρα να σε εξηγήσω τι είναι τα ειδικά τραβηκτικά δικαιώματα, αλλά ήταν ένα, ένα μέσο το οποίο χρησιμοποιήθηκε πολύ σε αυτή την κρίση. Εφόσον λοιπόν μιλήσετε για την Κένια, θα ήθελα να σας πω ότι ήταν πολύ σοβαρή η κατάστασή τους και εμείς ε, τους δανείσαμε. Ε, πώς ε, αυτό μπορεί να γίνει, μπορεί μέσω της παρεμβολής των G20 και το 2009 όχι μόνο οι γνωστές ε, χώρες αλλά και αναδιόμενες αγορές συνέβαλαν, αναδιόμενες χώρες και στο χάρτη εδώ που δεν θα δείτε για πολύ βλέπετε τα προγράμματα που έχουμε τώρα που λειτουργούν πολύ καλύτερα από τις προηγούμενες κρίσεις διότι βλέπουμε ότι υπάρχει μία πιο ομαλή ε, εξίσωση της πορείας και των αποτελεσμάτων. Βεβαίως ε, λέγεται ότι το ε, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο χρειάστηκε να αντιμετωπίσει την κρίση έχοντας πίσω του μια καλή περίοδο ε, αλλά θα μπορούσαμε βέβαια να έχουμε και καλύτερα αποθήματα. Δεν ήμασταν μόνοι. Ε, έπρεπε να ε, επικεντρωθούμε στις χρηματοοικονομικές αγορές, στις έγκαιρες προειδοποιήσεις και στην κάλυψη των ανισοτήτων. Και τώρα είμαστε στην ανάκαμψη. Εφέτος περιμένουμε 4% παγκόσμια ανάπτυξη και βέβαια όλα αυτά εξαρτώνται από την ε, ε, στήριξη της πολιτικής ε, και την επίλυση του προβλήματος του φορολογικού διότι βλέπετε ότι ιδίω στις αναπτυγμένες οικονομίες υπάρχει μία αύξηση του δανεισμού και των χρεών συγκεντρώσαμε λοιπόν το 2006 όλους τους ενδιαφερομένους. Το 2007 προσπαθήσαμε να συμφωνήσουμε πώς θα προσορμαζόντουσαν όλοι, αλλά μετά μας προέκυψε η κρίση και Έχω ένα έγγραφο που δεν υπάρχει στις διαφάνειες όπου βλέπετε τι κάναμε για να μειώσουμε τις παγκόσμιες ανισότητες και έχω μία προβολή για το 2014 όπου βλέπετε ότι θα υπάρχουν ακόμη ορισμένες ανισορροπίες διότι υπάρχουν ορισμένες χώρες όπου έχουν πλεόνασμα χρειάζεται να ενισχυθεί η εσωτερική ζήτηση και σε άλλες χώρες θα χρειαστεί να ενισχυθεί η προβολή προφορά, προσφορά είτε από τον δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Το ερώτημα είναι τώρα εάν έχουμε εστιαστεί στα προβλήματα του συστήματος και όχι τόσο πολύ στα διμερεί. Όσον αφορά την διακυβέρνηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου υπάρχει ένα πρόβλημα διότι πρέπει να υπάρξει μία μετακίνηση κατά 5% των ε, ποσοστώσεων προς τις ε, δυναμικά αναδυόμενες ε, χώρες Επίσης ε, βλέπετε ότι ε, σχετικά με τους G20 που ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής ε, υπάρχουν συνεδριάσεις μεταξύ των κρατών μελών υπάρχουν ισχυρά σημεία αλλά και αδυναμίες διότι ορισμένες χώρες είναι τελείως απούσες από αυτό το σύνολο. Και το τελευταίο θέμα που θα ήθελα να πω στο 1,5 λεπτό είναι ότι όσον αφορά τους κανόνες του παικτηριού για τις πληρωμές είναι ότι το καλό είναι ότι αντέξαμε την κρίση αλλά έχουμε και περιορισμούς. Δηλαδή ανέφερε και ο προηγούμενος ομιλητής για τις ροές του συστήματος διότι πολλές χώρες δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση της ρευστότητα όταν τη χρειάζονται, δεν υπάρχει ένα αυτόματο σύστημα και αυτό υπάρχει ε, πρόβλημα για ορισμένες χώρες σαν τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τις χώρες όπου υπάρχουν ε, μεγάλα αποθέματα ε, οι οποίες όμως δεν μπορούν να αντισταθμίσουν τις χώρες τις ελληματικές και εδώ βλέπετε ότι έχουμε μία συσσόρευση των αποθεμάτων τα οποία εκτινάσσονται και είναι ένα πρόβλημα που δημιούργησε το, δημιουργήθηκε στο Διεθνές Νομισματικό Σύστημα. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε λύσεις. Ε, καταρχήν όπως ε, ανέφερε ο προλαλής μέσω των ειδικών τραβηκτικών δικαιωμάτων και δεύτερον ε, εάν δεν βρείτε αλλού χρηματοδότηση μπορείτε να απευθυνθείτε σε μας. Ευχαριστώ. Αυτό ήταν θαυμάσιο. Και ερχόμαστε τώρα στον επόμενο ομιλητή. Ο Σάνικο Πό όμως το έχει το λόγο τώρα να μας παρουσιάσει τις ιδέες του. Σα ευχαριστώ πολύ. Μου ζητήθηκε να μιλήσω για τη διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών αγορών και πιστεύω πως ήταν ενδιαφέρον να αρχίσουμε με το ερώτημα της διαχείρισης από τις χρηματοπιστωτικέ αγορές. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε. Είναι μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην Σοβιετική Ένωση και τη Δύση ήταν ότι στη Σοβιετική Ένωση η κυβέρνηση καθόριζε τις τιμές. 24 εκατομμύρια τιμές για κάθε γραβάτα και για κάθε φρατζόλα ψωμί που πουλιόταν στα σούπερ μάρκετ. Στο δικό μας σύστημα οι αγορές καθορίζουν τις τιμές. Άρα λοιπόν οι αγορές είναι ένα πολύ σημαντικός μηχανισμός διακυβέρνησης. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για διακυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο σημαντικές είναι αυτές οι αγορές γιατί αυτές είναι που μας ε, διακυβερνούν. Επίσης είναι καλό να ξεκινήσουμε μια απλή ερώτηση, δηλαδή να πούμε τι είναι αυτές οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, λέει ότι οι αγορέ ε, ορίζουν, ε, λέει πόσο μπόνους πρέπει να πληρώσουν. Οι αγορές ορίζουν ότι το, το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο. είναι Επίσης αποφάσισαν ότι η το να χρηματοδοτηθούν υποθήκε, τα υπόθηκα δάνεια δανείζοντας ε, ε, στις αγορές που δεν δάνειζε κανένας άλλο ήταν πολύ καλύτερο από το να δίνονται ε, από την Northern, να δίνονται δάνεια σε αυτές τις αγορές παρότι η Northern Rock δεν το έκανε. Αυτές είναι οι αγορές που καθορίζουν ε, ποιες ε, ε, μετοχές αυξάνονται και ποιες πέφτουν. Δεν πρέπει να ξεχνάμε λοιπόν ποιες είναι αυτές οι αγορές, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε και ούτε και ποιος είναι ο κόσμος. Ο κόσμος είναι αυτός που συμβάλλει, στη... είναι και ο κόσμος που δικεί τις τράπεζες, οι τραπεζίτες, αλλά και οι traders υψηλή συχνότητα. Είναι πολύ σαφές ότι υπάρχουν πλονεκτήματα στη χρηματοπιστωτική αγορά και γι' αυτό και δούμε σε ευημερή κοινωνία υπάρχουν όμω και σαφεί περιορισμοί και θα πρέπει να υποθεί ότι σε αυτόν τον νέο κόσμο του 21ου αιώνα αυτοί οι περιορισμοί έχουν ε, αποκτήσει πολύ μεγαλύτερη σημασία και γι' αυτό και το θέμα είναι τόσο σημαντικό. Τι διαφέρει λοιπόν στον 21ο αιώνα. Ο κόσμος είναι πολύ πιο ε, λεξαρτημένο, ε, συνδέεται περισσότερο, υπάρχουν διασυνοριακέ ροέ εμπορίου, χρηματοδότηση, τρομοκρατία, οτι, οτιδήποτε κυκλοφορεί πιο γρήγορα. Οι μεταφορές, οι επικοινωνίες, οι τεχνολογικές πρόοδοι έχουν σημάνει πως τα πράγματα ρέουν ταχύτατα με πολύ ταχύ ρυθμα και είδαμε και την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας. Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Το πρώτο είναι γιατί παλιότερα οι τοπικές αποφάσεις είχαν τοπικό αντίκτυπο. Όμως λόγω αυτής της ε, διασύνδεσης οι τοπικές αποφάσεις που, γίνονται, που λαμβάνονται αυτή τη στιγμή πολύ συχνά έχουν παγκόσμιο αντίκτυπο. Ο βαθμός εξωτερικότητας ε, αλλά και οι μη ε, υπολογισμένες ο μη υπολογισμένο αντίκτυπο του άλλου έχουν ε, ε, αναταράξει ολόκληρο τον κόσμο. Ένα μικρό νησί τη Καραβική αποφασίζει να γίνει παράδεισο φορολογικό και ταυτόχρονα αυτό σημαίνει πω η γερμανική φορολογική κατάσταση κινδυνεύει. Έπειτα, ο ρυθμό τη ζωή έχει γίνει πολύ ταχύτερο. Δείτε, α πούμε, τι ταχύτητε των χρηματοπιστωτικών αγορών. Του τρέντερ υψηλή συχνότητα που εμπορεύονται 30.000 φορές μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Γιατί όλα αυτά είναι σημαντικά. Γιατί η εξωτερικότητα συνδέεται με τον αυξανόμενο ρυθμό της ε, ζωής. Αυτό σημαίνει ότι η απειλή της μετάδοσης, ε, η απειλή της μετάδοσης προβλημάτων που δημιουργούνται σε ένα κομμάτι του συστήματος και επηρεάζουν ένα άλλο κομμάτι, ε, πολλαπλασιαζόμενα εντωμεταξύ, είναι πολύ μεγαλύτερος. Παλιότερα η κίνδυνη ήταν τοπική, τώρα η κίνδυνη είναι συστημική και οι υπάρχοντες ε, μηχανισμοί διακυβέρνηση που έχουμε, τα παγκόσμια, τα διεθνή ιδρύματα ή και τα εθνικά ιδρύματα, είναι, δεν είναι σε θέση να χειριστούν τόσο περίπλοκα συστήματα και κοινοτομίες. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι ένα νέο σύστημα και θα επανέλθουμε σε αυτό, ελπίζω προς το τέλος. Ας πούμε επίσης ε, για τις αγορές. Αυτό που είναι πολύ, καλά, πολύ γνωστό σχετικά με τις αγορές είναι πως είναι φοβερές στην να χειριστούν την εξωτερικότητα. Δηλαδή δεν ασχολούνται με την ε, ρήπανση που κάποιο παράγοντας μπορεί να προκαλέσει με τα μεταδοτικότητα. Οι κυβερνήσει πρέπει να το πράξουν αυτό. Έπειτα οι αγορέ δεν μπορούν να παρακολουθήσουν το συστημικό κίνδυνο τακτικά, να τον εποπτέψουν. Αυτά είναι δύο χαρακτηριστικά των αγορών και γι' αυτό στον 21ο αιώνα οι αγορέ θα ε, δυσκολευτούν περισσότερο για να παίξουν το ρόλο δημιουργία αξία που έπαιξαν στο παρελθόν. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι η ε, οι αγορές ε, προσανατολίζονται περισσότερο στα κέρδη. Αν δούμε τις εταιρείες του Dow Jones, αναφέρουν οι περισσότερες κέρδη που είναι δύο παραπάνω cents από τις προβλέψεις των ε, διευθυντών τους. Οι περισσότεροι τους ζητήθηκαν να, ε, να τους ζητήθηκε μάλλον να επιλέξουν μια επένδυση και ανάλογα με το, το κέρδος που τους δώσει, περισσότερο επιλέγουν τις επενδύσεις που μακροπρόθεσμα καταστρέφουν την αξία. Άρα λοιπόν, Έχουμε κάποιον στον κόσμο που να είναι σε θέση να χειριστεί τις προκλήσεις διαχείρισης διακυβέρνησης του 21ου αιώνα. Όχι ακόμα και γι' αυτό πρέπει προς αυτό να προχωρήσουμε. Για να μιλήσουμε για την οικονομία πιο συγκεκριμένα. Αν πάμε στη δεκαετία του 50, όπου εγώ δεν είχα ακόμα γεννηθεί, οι τιμές του χρηματιστηρίου υπολογίζονταν από τους, τα, τους μικρούς υπολογιστές χειρός. Οι επενδυτικές τράπεζες δεν μπορούσαν να είναι εμπορικές τράπεζες και τα κίνητρα καθώς και οι ρυθμιστικές δομές ήταν κατακαιρματισμένες σε ολόκληρο τον κόσμο. Τα διάφορα κομμάτια του κόσμου είχαν διαφορετικές ρυθμιστικές δομές. Αν τώρα έρθουμε στη σημερινή ημερομηνία, κάθε φορέα της αγοράς έχει άμεσα πρόσβαση στις τιμές της αγοράς σε ολόκληρη την παγκόσμια αγορά ε, ε, οι έλεγχοι των κεφαλαίων έχουν ε, καταργηθεί, η απορρίθμιση σήμαινε πως δεν υπήρχε πλέον χωριστά επενδυτικές τράπεζες και εμπορικές τράπεζες, οπότε σε τι καταλήξαμε. Σκεφτείτε τα, τη θεωρία των χαρτοφυλακίων. Η ιδέα είναι αυτό που θα έλεγε και η γιαγιά μας, δηλαδή μην βάζεις όλο το αυγά στο ίδιο καλάθι. Σημαίνει δηλαδή πως τουλάχιστον αν, χαλά, αν ζημιωθεί ένα καλά δεν θα χάσει όλο το αυγά. Δηλαδή προσπαθείς να βάζεις αυγά σε διάφορα καλάθια. Αυτή ήταν η ιδέα του χαρτοφυλακίου. Και αυτό εντάξει το 50 λειτουργούσε γιατί υπήρχαν ένα σωρό καλάθια. Μα τώρα όμως κάθε συγκεκριμένος ε, φορέας προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την διαφοροποίηση, πράγμα που είναι λογικό και για αυτούς. Αυτό λέει και ο, λένε και οι ρυθμιστές, αυτό λέει και η θεωρία και τελικά εκτίθενται στους κινδύνους όλων των αγορών σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτό σημαίνει πως η επιδίωξη της διαφοροποίησης ε, που οδηγήθηκε στο άκρο της οδήγησε σε ομοιομορφία. Σχεδόν όλοι οι μεγαλύτεροι οικονομικοί φορείς ε, στην, ε, στον κόσμο επενδύουν σε παρόμοια χαρτοφυλάκια και γι' αυτό το σύστημα είναι εξαιρετικά έθραυστο. Η διαφορά είναι πως κανένα συγκεκριμένο ίδρυμα δεν είναι τόσο εύθραυστο όσο ήταν παλιότερα, αλλά το σύστημα ολόκληρο είναι. Και αυτό που συνέβη είναι ακριβώ μια απλή απόδειξη αυτή τη τάση. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Τα διδάγματα είναι σαφή για τη διακυβέρνηση και για τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Το πιο σημαντικό είναι πως υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά προβλήματα κινήτρων. Αν δούμε τα κέρδη των τραπεζών, οι τράπεζες παλιά είχαν ε, την, το ίδιο πλεόνασμα 5 με 10% όπως η πραγματική οικονομία. Και έπειτα κάτι συνέβη τη δεκαετία του 70 και την τελευταία δεκαετία είχαμε απόδοση 25% σε σε χρεόγραφα. Ε, και γιατί γινόταν όλο ένα και περισσότερο μόχλευση. Και όλοι όσοι γνωρίζουμε κάτι από χρηματιστήρια ξέρουμε ότι όσο περισσότερο κέρδο, ε, ε μάλλον ρίσκο παίρνεις, τόσο περισσότερο κέρδος μπορεί να έχεις, αλλά και τόσο και μεγαλύτερο κίνδυνο. Άρα λοιπόν αυτό προσπάθησαν να διευρύνουν και να αυξήσουν τη μόχλευση στο σύστημα. Και ακριβώς αυτό συνέβη. Αυτές οι δομές κινήτρων είναι πολύ σημαντικές για να δούμε πώς ε, λειτουργούν τι ρόλο παίζουν οι αγορές. Οι αγορές και οι φορείς της αγοράς θα δείχνουν ότι θα πρέπει να είναι όλα αυτά σε σχέση με την πραγματική οικονομία, να είναι υπόλογοι στην πραγματική οικονομία και όχι μόνο στους όρους της αγοράς, γιατί πολλές, πολλοί από τους κανονισμούς που είχαμε βασίζονταν ε, στην χρήση των τιμών της αγοράς για να, για να ζυγίζουν το κίνδυνο. Αλλά δεν λειτουργήσε αυτό όπως έπρεπε. Γι' αυτό και λοιπόν η λύση μπορεί να είναι η εξή. Είτε να επανέλθουμε σε ένα κατακαιρματισμένο σύστημα το οποίο να είναι διαφοροποιημένο και είναι αποκομμένο το ένα από το ΔΕΗ ή θα μπορούσαμε να καταλήξουμε σε ένα παγκόσμιο σύστημα που πραγματικά θα χειριστεί το κενό διακυβέρνησης, δηλαδή δομημένα σώματα, ή ε, οργανισμοί που θα είναι ευλίγιστα και θα, και θα μπορούν ε, να κινηθούν πολύ γρήγορα. Δεν μοιάζουν τίποτα με αυτό που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Uh,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 Θα σας ε, παρουσιάσω μία συγκεκριμένη πρόταση, δηλαδή ε, μία ιδέα για μία γενική, ένα γενικό φόρο για τις δημοσιονομικές ε, συναλλαγές. Και αν κοιτάξουμε τον, τη μεταπολεμική περίοδο, βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο περίοδοι. Καταρχήν η ευημερία ε, μέχρι το 1970 με μία συνεχή εξέλιξη του κοινωνικού κράτους και μετά 30 χρόνια με ε, δανεισμό του κράτους με κοινωνικές ανισορροπίες και ε, συνεχώς επιδεινωμένη κατάσταση. Η προσπάθεια κέρδους είναι η βασική η κινητήριος δύναμης του καπιταλισμού και στην πρώτη ε, περίοδο αναφέρθηκε ε, σε ορισμένα στοιχεία τα οποία ανέφερε ο πρώτος ομιλητής, ο κύριος Παντώα Σιώπα, ε, χαμηλές, χαμηλά επιτόκητα, σταθερές τιμές, ενώ στη δεύτερη περίοδο μιλάνε μόνο για να αφήσει κανείς τα χρήματά του να δουλεύουν. Δηλαδή υπάρχει, υπήρχε στην αρχή ένας ρεαλιστικός καπιταλισμός και στη δεύτερη περίοδο ένας δημοσιονομικός καπιταλισμός και αν δείτε τη δεύτερη περίοδο βλέπετε ότι υπάρχει ένας ε, αναπτυξιακός κύκλος αλλά ε, στο προηγούμενο κύκλο φτάσαμε στην ε, κρίση του 1930 η οποία ήταν ριζική ε, και από εκεί δημιουργήθηκε ένα διαφορετικό καπιταλιστικό σύστημα με συνδυασμό των συμφερόντων του, του πραγματικού κεφαλαίου και της εργασίας ε, κατά του δημοσιονομικού κεφαλαίου. Αυτό ε, βλέπουμε σε μία σχέση μεταξύ ε, του πραγματικού κεφαλαίου και της εργασίας και τώρα βρισκόμαστε σε μία νέα μεταβατική κρίση όπου πάλι από τον δημοσιονομικό καπιταλισμό θα επανέλθουμε σε σχέσεις ε, ε, ρεαλιστικού καπιταλισμού. Πώς μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τα χαρακτηριστικά αυτών των τάσεων. Ε, καταρχήν βλέπουμε τις ισοτιμίες, τις τιμές των πρώτων υλών, την ε, αξιοποίηση της αγοράς, τη σχέση των επιτοκίων με το ποσοστό αυξήσεως και την ε, σχέση μεταξύ πραγματικών ε, και εικονικών συναλλαγών. Εδώ βλέπετε ε, την ακολουθίες του της ανωδικής αγοράς και της πτωτικής αγοράς, bull market και bear market, από το 1960 μέχρι το 2000 μετά υπάρχει μια νέα διακύμανση μετά το 2000 και μετά καταραίει και πάλι. Ε, παραδείγματος χάρη η ε, τιμή συναλλάγματος του ευρώ πάλι έχει ε, μεγάλες διακυμάνσεις, χάνει το 1 τρίτο της τιμής συναλλάγματός του, μετά τη διπλασιάζει. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω τι σημαίνουν αυτές οι διακυμάνσεις. Βλέπουμε όμως δύο γραμμές και η μαύρη γραμμή είναι οι λανθάνουσες τάσεις, δηλαδή δηλαδή οι ε, μετακινήσεις των, των τιμών των περιουσιακών στοιχείων και ε, της κερδοσκοπίας η οποία χρησιμοποιείται σε διάφορες συχνότητες βλέπετε εδώ σε πέντε λεπτά τις διακυμάνσεις της ε, τιμής συναλλάγματος δολαρίου ε, εναντί ευρώ σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία και έχετε ακούσει για τα trade following hedge fund, hedge funds, δηλαδή πρόκειται για συστήματα τα οποία ενισχύουν αυτές τις τάσεις. Άρα, εάν κοιτάξει κανείς την τελείως βράχη πρόθεσμη συμπεριφορά των συναλλαγών είναι ότι οι μακροπρόθεσμες ε, τάσεις είτε των μετοχών, είτε των τιμών συναλλάγματος ή των πρώτων υλών δεν είναι παρά μία συσσόρευση μικροσυναλλαγών πενταλέπτων, τριλέπτων επί σειρά ετών. Εάν δηλαδή συσσωρεύσει κανείς όλες αυτές τις διακοιμώσεις και αν μπορεί να τις μειώσει θα μπορούσε να καταπολεμήσει και την μακροπρόθεσμη αστάθεια και και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ τις αυξομοιώσεις ε, της τιμής ε, του πετρελαίου και βλέπετε ότι αυτό εδώ είναι οι πιο ελεύθερες αγορές οι οποίες και πάλι δίνουν λαθασμένα, λαθασμένες ενδείξεις σχετικά με τις τιμές. Και ε, είναι μία πολύ αργή διαδικασία ε, όπως είδαμε και στην προηγούμενη οικονομική κρίση. Δηλαδή χρειάστηκαν ε, πολλά χρόνια για να μπορέσουν να προσαρμοστούν οι δημόσιες οικονομίες. Είπα όμως ότι οι μακροπρόθεσμες διακοιμάνσεις των πιο βασικών ε, σημείων του δολαρίου παραδείγματος χάρη στην κόκκινη γραμμή η οποία έχει τέτοιες τεράστιες διακοιμάνσεις αποσταθεροποιεί την παγκόσμια οικονομία διότι η τιμή του πετρελαίου αντέδρασε με δύο πετρελαϊκές κρίσεις. Δεν αντιληφθήκαμε τότε ότι το σοκ της τιμής του πετρελαίου ήταν μία απάντηση στις διακυμάνσεις και υποτιμήσεις του νομίσματος το οποίο ε, τιμάτο το πετρέλαιο. Εδώ βλέπουμε καταρχήν τη σχέση μεταξύ της ε, ε, πορείας ε, του, της ισοτιμίας του δολαρίου και ε, βλέπετε ότι δεν υπήρχε ε, επίσης ε, σχετικά με την ανάπτυξη της παγκοσμίου αγοράς μία ύφεση επί πολλά χρόνια. Στο τέλος της δεκαετίας του 50 είχαμε πλήρη απασχόληση και μία βασική προϋπόθεση στο κάτω διάγραμμα είναι ότι ε, τα επιτόκια ήταν χαμηλότερα από το ε, ποσοστό αναπτύξεως, άρα ε, είναι ακόμη ένα παράδειγμα για αυτό που σας ονόμασα ως ρεαλιστικό καπιταλισμό. Η κατάσταση δεν είναι πλέον ανεκτή όταν οι non-financial ε, business, δηλαδή οι μη δημοσιονομικές ε, επιχειρήσει δημιουργούν ε, περισσότερο κεφάλαιο από ότι ουσιαστικά είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή όταν σας λένε αφήνετε το κεφάλαιό σας να δουλεύει, ε, και προχωρούν δημοσιονομικά δεν, ε, δεν μπορεί κανείς ε, να προχωρήσει σωστά και βλέπετε εδώ σε αυτό το διάγραμμα σας είπα ότι ένα βασικό στοιχείο είναι η τελεία ε, έλλειψη συντονισμού μεταξύ πραγματικών αγορών και αγορών πρώτων υλών. Εδώ βλέπετε ότι ε, ο παγκόσμιο ΑΕΠ αντικατοπτρίζεται στο οχταπλούν στις ε, συναλλαγές της διεθνής, δηλαδή αυτό οφείλεται στα παράγωγα ε, τα χρηματιστηριακά τα οποία διακινούνται στις αγορές από κερδοσκόπους. Και εδώ θα συνδέσω αυτά που είπα με την τελική παρατήρηση. Δηλαδή, αν όντως μακροπροθέσμος υπάρχει μία υπέρβαση των τιμών στο, ανά τον κόσμο, και ε, υπάρχει μία συσσόρευση μικρών διακοιμάσεων τότε ε, η κερδοσκοπία αυτή βραχυπρόθεσμα γίνεται πιο δαπανηρή και γενικοποιεί την ε, αρχη καιν στομπιν, δηλαδή όλες οι δημοσιονομικές ε, συναλλαγές θα πρέπει να έχουν μία ενιαία φορολόγηση 0,1%, 0,05% και η πρότασή μας θα εξασφάλιζε ότι με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο ε, θα επιβαρυνθούν μόνο οι συναλλαγές οι οποίες είναι πολύ βραχυπρόθεσμα με μεγάλο leverage, με μεγάλη εγγύηση, μόχλευση. Δηλαδή ε, θα πληρώνετε τότε 0,05 cents, δηλαδή ένα πολύ χαμηλό ποσό. Όλα αυτά δεν μπορούν καν να εμφανιστούν ε, στο κομπιούτερ και βλέπουμε ότι ε, για την Ευρώπη με 0,05% θα μπορούσε κανείς να καταλήξει σε ε, μία πρόσοδο 350 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστώ. Ε, ξέρω ε, ότι εδώ έχουμε περιορισμένο χρόνο, οπότε δίνω μέσω το λόγο στον πρώτο ο οποίος το ζήτησε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο που καταρτίζω αυτή τη στιγμή και θα με βοηθήσει η δημόσια κρόση αφορά και την παγκόσμια διακυβέρνηση, τις παγκόσμιες ανισορροπίες. Οπότε οι ερωτήσεις μου... Έχω ερωτήσει προς τον κύριο Μπέρτ Βανσέλμ. Οι παγκόσμιες ανισορροπίες ε, συνετέλεσαν στην τρέχουσα χρηματοπιστωτική κρίση, ε, κρατώντας χαμηλά τα επιτόκια και ενισχύοντας την ε, απληστία για μεγάλες αποδόσεις. Αυτό που έδειξε είναι ότι η διαχείριση δεν ήταν σωστή, γιατί οδήγησε σε φούσκες. Οπότε το επίπεδο δημόσιο χρέους σε πολλές περιπτώσεις δεν μας επέτρεψε να απορροφήσουμε μεγάλα φορολογικά ανάβσματα. Και έχω διτή ερώτηση. Καταρχήν, πιστεύω ότι θα πρέπει να μειώσουμε τα κριτήρια του Μάστριχτ από το 6% από το 60% στο 50% ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το παρέτητο πακέτο φορολογικών εναυσμάτων. Στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο συντάξατε μια πολύ σημαντική έκθεση που αμφισβήτησε τον μακροπρόθεσμο ποσοστό πληθωρισμού του 2%. Μπορείτε να μας το σχολιάσετε ένα στόχος πληθωρισμού 2% θα επιτρέψει την απορρόφηση κραδασμών ε, από το σύστημα σε μια περίοδο κρίσης. Για την πρώτη σας ερώτηση, σε ό,τι αφορά τα κριτήρια του Μάστριχτ και την ε, χαλάρωσή τους, μάλλον είναι ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση παρά προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Πάντως, ε, έχουμε μέσους όρους για το 2014 που είναι, οι προβολές που κάνουμε είναι γύρω στα 110%. Οπότε είτε 50-60% είναι πολύ χαμηλότερο ποσοστό από τις προβολές που κάνουμε για τις αναμενόμενες ε, αναλογίες του χρέους ως προς το ΑΕΠ. Σε ό,τι αφορά την διαδικασία αξιολόγησης δεν πρόλαβα να την αναπτύξω. Πάντως υπάρχουν ελπίδες ότι θα οδηγήσει σε κάτι. Ε, όπως είπα, προσπαθούμε το, προσπαθήσαμε το 2006 και 2007 στις πολυμερείς διαπραγματεύσεις, αλλά η διαφορά σήμερα είναι ότι το πρόγραμμα του G20 για την αμοιβαία αξιολόγηση είναι του G20, δεν το διαχειρίζεται το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο. Πάντως ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από προηγούμενα εγχειρήματα με τον ίδιο σκοπό. Και την τρίτη σας ερώτηση για το έγγραφο et Τόλ. Αυτή η θέση δεν είναι η θέση, η επίσημη θέση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αναφέρεται σε ένα σημείωμα. Και αυτό που διέρευσε στον τύπο, ή μάλλον αυτό που κυκλοφόρησε στον τύπο, είναι ότι ε, η έκθεση Blanchard προβλέπει ότι είναι προτιμότερο πληθωρισμός 4% από τη 2%. Είναι, υπάρχει πολύ ενδιαφέρον έγγραφο για την ε, επαναπροσδιορισμό της μακροοικονομικής πολιτικής. Πολύ χρήσιμο αυτό το έγγραφο και νομίζω ότι είναι υπεραπλουστευτικό από ολόκληρο αυτό το έγγραφο να μένουμε μόνο σε, ένα, μια πρόταση του στόχου του 2% για τον πληθωρισμό. Ο Χέλμουντ Σμιθ είχε πει 6% ε, πληθωρισμός είναι προτιμότερος από το 6% ενεργεία, είχε πει ο πρώην καγκελάριος Χέλμουντ Σμιτ. Δανούτα Χιούμπλερ. Ευχαριστώ. Όλοι σας μιλήσατε για την κρίση με όριστο χρόνο, σαν να έχει περάσει και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό. Φαίνεται να περνάμε σε μια πιο ομαλή κατάσταση μετά την έξοδο από την κρίση. Βέβαια έχουμε πιο αργούς ρυθμούς ανάπτυξης, ε, μια εσωστρέφεια από πολλές χώρες και χρειαζόμαστε μια παγκόσμια διακυβέρνηση και περισσότερο ρυθμισμένα χρηματοπιστωτικά συστήματα. Βέβαια δεν είναι σαφές τι γίνεται με το δημόσιο χρέος, γιατί εκεί υπάρχει κίνδυνος να πέσουμε σε μια παγίδα με το δημόσιο χρέος και να καταλήξουμε σε μια κρίση δημοσίου χρέους. Έχω μια ερώτηση για να σχολιάσετε. Η αποκατάσταση της δημοσιονομικής ισορροπίας χωρίς ε, να διακυβεύσουμε τα επίπεδα τιμών στις αναπτυσσόμενες χώρες και γενικώ είναι τεράστια πρόκληση. Ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει να έχει ένα σχέδιο για να αποκαταστήσει την δημοσιονομική ισορροπία χωρίς ταυτόχρονα να ενδώσει τον πληθωρισμό. Ποιος θέλετε να απαντήσει στην ερώτησή σας. Όποιος να είναι. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που θα πρέπει να έχουμε υπόψη είναι ότι η γη δεν είναι χρεωμένη στον Άρη. Είναι θέμα κατανομής. Όταν μιλούμε λοιπόν για το δημόσιο χρέος, κάποιος ε, χρωστάει χρήματα σε άλλον. Οπότε αυτό είναι ένας απλός τρόπος να αντιμετωπίσουμε την κρίση του δημόσιου χρέους. Αν κάποιος ρώτανε από τον πλανήτη Άρη και έλεγε θα κάνουμε διαφορετική κατανομή και θα υπάρξουν ζημίες. Ναι, αλλά τώρα με τις τράπεζες δεν έγινε κάτι τέτοιο. Εκεί οι δανειστές δεν ανέλαβαν τις ζημιές, τις ζημιές τις ανέλαβαν οι κυβερνήσεις. Γι' αυτό δημιουργήθηκαν ε, δημοσιονομικές ανισορροπίες. Υπάρχουν τρεις πιθανοί τρόποι προσέγγισης. Καταρχήν, θα πρέπει να αυξήσουμε το φορολογικό εισόδημα, τα φορολογικά έσοδα. Με αυτό το στόχο συμφωνούμε όχι, όλοι, ότι για να αυξήσουμε τα φορολογικά έσοδα θα πρέπει να περιορίσουμε την φοροδιαφυγή ή τη φοροαποφυγή. Μέσω του G20 έγιναν κάποιες ε, προτάσεις για ανταλλαγή πληροφοριών φορολογικών, αλλά αυτέ είναι διμερεί συμφωνίε. Αν όλε οι χώρε είχαν τέτοιε διμερεί συμφωνίε μεταξύ του, θα χρειαζόμασταν 18.000 ε, και τέτοιε συμφωνίε. Και έχουμε 3.000 και. Και συνάπτουμε συμφωνίε ε, με το ρυθμό 10 το χρόνο. Θέλουμε επιγόντω μία πολυμερή συμφωνία για ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων. Να να αναχθεί σε πολυμερές επίπεδο ε, μία φορολογική συμφωνία του ΩΣΑ ή κάποιες αντίστοιχες προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και να μην περιοριστούν σε διμερείς συμφωνίες. Και με τους φορολογικούς παραδείσους ε, γίνεται μία μετάβαση προς τα έξω του προβλήματος του φορολογικού. Επίσης, ε, το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο είχε κάνει μία πρόταση. Εγώ όταν ασχολόμουν με τις αναπτυσσόμενες χώρες, τους ε, υποδεικνύαμε να έχουν έναν ε, υγιή μηχανισμό δημόσιου χρέους, γιατί πολλές φορές δεν μπορούσαν να αποπληρώσουν το χρέος τους και η Ευρώπη τότε αδιαφορούσε γιατί το πρόβλημα ήταν ε, αλλού. Ήταν στην Νότια Αφρική, στην Δυτική Σαχάρα. Τώρα όμως η Βραζιλία δεν έχει χρέος, η Ευρώπη είναι που έχει τα δημόσια χρέη. Είτε τώρα πάντως είτε στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε ένα συστηματικό προβλέψιμο τρόπο για να αντιμετωπίσουμε το δημόσιο χρέος και το κεφάλαιο 9 του, του μοντέλου, γιατί το χρέος των κοινοτήτων είναι πολύ καλό υπόδειγμα. Γιατί τα πρώτα έσοδα πηγαίνουν στην απασχόληση, στην υγεία, στην παιδεία και μόνο όταν αν περισσεύσουν κονδύλια δίνω, επιστρέφονται στους θενιστές. Ίσως αυτό το υπόδειγμα θα μπορούσαν να το ακολουθήσουν και άλλοι. Θα πρέπει επίσης να βρεθούν και νέες μορφές φορολογικών εσόδων. Ο Στέφαν μίλησε για τον φόρο των διεθνών χρηματοπιστωτικών συναλλαγών ή κάποιων άλλων εισφορών από τις τράπεζες. Αν εξετάσουμε τι αντίκτυπο έχουν οι φόροι αυτοί στην ανάπτυξη. Για παράδειγμα, πολλέ φορέ χρηματοδοτούνται κάποια φιλοπεριβαλλοντικά σχέδια, η αύξηση τη απασχόληση ή το, η μείωση του εργατικού κόστου. Αυτοί οι φόροι είναι φόροι για τον εξωτερικό χαρακτήρα που μειώνουν τις, τα ελλείμματα. Υπάρχει λοιπόν τρόπο να αντιμετωπίσουμε μακροπρόθεσμα το δημόσιο χρέο, αλλά πρέπει να υπάρξει συντονισμό. Ο κύριο Σουλμάιστερ. Μία σύντομη απάντηση τα ελλείμματα και τα πλεονάσματα είναι αλληλοεξαρτούμενα. Δεν έχει νόημα να σκεφτόμαστε το έλλειμμα χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι κάπου αλλού υπάρχει πλεόνασμα. Στην άλλη πλευρά υπάρχει πλεόνασμα, είναι άλλη όψη. Ο Dr. Κέινς ασχολήθηκε με το θέμα αυτό όταν ετοιμαζόταν για τον Bretton Woods στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ήταν εξοικειωμένο με μια γενική λύση που έχει τα εξή χαρακτηριστικά. Αν μια χώρα έχει έλλειμμα, είτε στις εξωτερικές σχέσεις, είτε στις εσωτερικές, έλλειμμα του προπολογισμού, η συνταγή είναι πάντα η χώρα αυτή με το έλλειμμα ή ο τομέας με το έλλειμμα να μειώνει τις δαπάνε του. Ο Κέινς επιχειρηματολόγησε ότι από συστημική άποψη αυτό σημαίνει κατά ανάγκη ότι η διαδικασία προσαρμογής συνοδεύεται από μία μείωση της οικονομικής δραστηριότητας. Γιατί ο τομέας με το έλλειμμα μειώνει τις δαπάνες και ο τομέας με το πλεόνασμα δεν κάνει τίποτα. Οπότε η δική του συμβουλή είναι δεν είναι καλύτερο να ζητήσουμε από τον τομέα που έχει πλεόνασμα να αυξήσει τις δαπάνες. Για παράδειγμα, Γερμανία και νότιότερες, νότιες χώρες όλοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι χώρες, όπως, χώρες του Νότου όπως η Ελλάδα, αλλά και η Ισπανία και η Ιταλία και η Πορτογαλία θα μειώσουν τις δαπάνες τους. Ποιος όμως θα πληγεί περισσότερα από μια τέτοια μείωση δαπανών? Πρώτα απ' όλα η Γερμανία, η χώρα που έχει το πλεόνασμα. Γιατί μέχρι στιγμή η Γερμανία είχε μαζικέ εξαγωγέ προ τι χώρε του Νότου. Αν τώρα και όλε αυτέ οι χώρε ταυτόχρονα μειώσουν τη ζήτησή του εξαιτία μείωση των δαπανών, η χώρα που θα πληγεί πρώτα απ' όλα είναι η Γερμανία. Θεωρητικά βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα το πλεόνασμα, η χώρα που έχει το πλεόνασμα να αυξήσει τις δαπάνες της. Και το ίδιο ισχύει για την εξομάλυση των δημοσιονομικών. Αν στην Ευρώπη όλες οι χώρες αρχίσουν από το χρόνο να μειώνουν συστηματικά τις δαπάνες τους, τότε θα περάσουμε στη δεύτερη φάση της κρίσης. Γιατί είπατε ότι όλοι είμαστε αισιόδοξοι. Σας είπα ότι βρισκόμαστε στην αρχή τώρα της κρίσης, όχι στο τέλος της κρίσης. Και η αρχή της κρίσης σημαίνει ότι στην επόμενη φάση οι συλλογικές αποταμιεύσεις των κυβερνήσεων εκτός από την αύξηση της απασχόλησης, μπορούν να οδηγήσουν και σε τη αύξηση της ανεργίας, μπορούν να οδηγήσουν και σε νέα ύφεση. Αυτά είναι απλά πράγματα στη μακροοικονομική θεωρία. Υπερβάως. Ευχαριστώ. Κύριε Σουλμάιστερ, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Καταρχήν ευχαριστώ για την ανάλυση σας για τους κύκλους του καπιταλισμού και είπατε για τη διαφορά τη ρήξη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και μάλιστα με την εξαφάνιση της γενιάς που γνώρισε την κρίση, που έζησε την κρίση του 29. Νομίζω εκεί υπάρχει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσαμε να περιλάβουμε στο συλλογισμό μας. Τώρα σε ό,τι αφορά την πρόταση για το φόρο των, των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, το γενικό φόρο αν ε, η καταπληκτική αυτή ιδέα δεν περάσει στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, έχει νόημα να την εφαρμόσουμε εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Κύριε Βανσέλμ, τι προτείνετε για τους φορολογικούς παραδείσους. Γιατί ό,τι θέλουμε μπορούμε να κάνουμε. Αλλά αρκούν τα συμπεράσματα του G20 ή ήταν μόνο μία φήμη που διαδόθηκε κάποια στιγμή. γιατί δεν είμαι σίγουρη ότι θα σημειώσουμε πρόοδο εκεί. Γιατί έγιναν τόσα σεμινάρια για τις ανισορροπίες που υπάρχουν διεθνώς, αλλά το αποτέλεσμα είναι μηδέν. Άκουσα αμέσως μετά την, το ξέσπασμα της κρίσης τον Κόρτον Μπράουν, τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, να τάσσεται υπέρ ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης. Εκεί όμως είχαμε τον προσδιορισμό των ε, παγκόσμιων ανισορροπιών. Τι νόημα έχει, τι χαρακτηριστικά θα μπορούσε να έχει ένα σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και κάτι άλλο συναφές. Πώς μπορούμε να παρεύουμε όταν εντοπίζουμε μια τέτοια φούσκα και ποιος ε, νομοποιείται να παρέμβει, ο νομοθέτης και ποιος θα προειδοποιήσει τον νομοθέτη ή οι κεντρικές τράπεζες. Καλύτερα φυσικά ο παγκόσμιος αυτός φόρος για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές να ισχύει, να ισχύει διεθνώς αλλά οι συναλλαγέ στις χρηματοπιστωτικές αλλαγέ γίνονται σε τρεις χρονικές ζώνες. Ανατολική Ασία, Ευρώπη και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Στην ευρωπαϊκή ζώνη των συναλλαγών δεν υπάρχει ανταγωνιστική αγορά. Και για να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Οι περισσότερες χρηματοπιστωτικές αλλαγέ γίνονται με συναλλαγές στα παράγωγα, στα παράγωγα προϊόντα. Όλες οι συναλλαγές σε παράγωγα στην Ευρώπη γίνονται μόνο σε δύο, ε, ε, δύο γίνονται στο Λονδίνο και στη Φραγκφούρτη, σε δύο χρηματιστήρια. Αν λοιπόν ε, θεσπίσετε έναν ε, χαμηλό φόρο συναλλαγών, Αποκλείεται αυτά τα δύο χρηματοπιστωτικά κέντρα να συμφωνήσουν, γιατί στις Ηνωμένε Πολιτείες έχουμε το Atlantic City και το Las Vegas. Εκεί γίνονται τα περισσότερα στοιχήματα. Και εκεί έχουμε εξωτερική μεταφορά, εξωτερικότητα και όλοι πηγαίνουν εκεί αν θέλουν να στοιχηματίσουν. Εκεί γίνεται όλος ε, ο τζόγος. Αλλά δεν υπάρχει, κατά τη γνώμη μου, συγκεκριμένος κίνδυνος αυτές οι αγορές να μετατοπιστούν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κίνδυνος να μεταγκατασταθούν. Για τις καθολικές ανισορροπίες αυτό είναι πολύ σημαντικό και είναι και το επίκεντρο της σημερινής συζήτησης. Ο πρώτος ομιλητής είπε ότι υπάρχει πρόβλημα γιατί η πίεση είναι πιο εμφανή σε ορισμένους ε, φορείς και από ό,τι σε άλλους. Οι για παράδειγμα, χρηματοδοτούν το χρέος τους με το ίδιο του το νόμισμα. Και μόνο για τις Ηνωμένες ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και χώρες που έχουν πλεόνασμα, που διαχειρίζονται τα πλεονάσματά τους και αποθυσαυρίζουν, συσσωρεύουν πόρους και αποθέματα. Νομίζω ότι υπάρχει μία σωστή συμβολή, συμβολή που, είναι, που ισχύει για όλους. Άλλοι την εφαρμόζουν και άλλοι χρειάζονται δάνειο. Γίνεται διάλογος και καταλήγουμε σε μία συμφωνία. Το θέμα είναι η διαδικασία προσαρμογής να γίνει παγκοσμίω, παγκοσμίως πιο ισορροπημένη. Γι' αυτό και αναφέρω τη διαδικασία του, της αξιολόγηση αξιολόγησης στο G20. Στην κρίση υπήρξε μεγάλο πνεύμα διεθνού συνεργασία και όλοι συνειδητοποίησαν ότι χρειάζεται συνεργασία για να εξέλθουμε από την κρίση. Και ανέφερε την απόφαση του Απριλίου του 2009 των G20 για τον τριπλασιασμό των πόρων του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Και αυτό στις αγορές είχε τεράστιο αντίκτυπο. Αυτή την ε, όθηση θα πρέπει να την εκμεταλλευτούμε. Γιατί όλοι είδαν ποια είναι τα καλά της συνεργασίας στην παγκόσμια οικονομία. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα μέσω της διαδικασίας αμοιβαίας αξιολόγησης του G20. Ουδέν σχόλιο για τους φορολογικούς παραδείσους. Δύο λόγια για τους φορολογικούς παραδείσους. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι οι σκανδιναβικές χώρες άρχισαν τη συνεργασία τους το 2006 και από κοινού διαπραγματεύτηκαν διμερείς φορολογικές συνθήκες. Γιατί λοιπόν να μην διαπραγματευτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τέτοιες φορολογικές συνθήκες εκ μέρους των κρατών μερών, ακόμη και αν γίνονται διμερός. Θα έχει και μεγαλύτερο διαπραγματευτικό βάρος. Είμαστε μεγαλύτερη οικονομία, σημαντικότερη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να προσφύγουν νομικά κατά του UBS και ζητούν ε, πληροφορίες για τις ε, αμερικανικές επενδύσεις στην Ελλοδαπή. εμείς είμαστε μεγαλύτερη οικονομία. Από αυτή την άποψη έχουμε πολύ μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ που την αφήνουμε αναξιοποίητη. Υπάρχει ένας, ένα σύστημα προαγγραφής ε, για τους φόρους. Ακόμη και η Αυστραλία έχει κάτι αντίστοιχα αρχεία για τους φορολογικούς παραδείσους. Μπορούμε λοιπόν να ασχοληθούμε με τη φοροδιαφυγή, αλλά δεν έχουμε στην Ευρώπη κάτι αντίστοιχο. Η συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να φέρει πολλούς καρπούς, χωρίς καν να χρειάζεται παγκόσμια συμφωνία και θα μπορούσαμε να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή. Και η κρίση μας έχει δείξει πόσο κατεπίγουσα είναι αυτή η αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ε, Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της φορολογίας των συναλλαγών γιατί είπατε ότι αυτό θα μπορούσε να αποκομίσει περίπου 300 δισεκατομμύρια ευρώ βασίζεται ε, ο υπολογισμός σας σε ένα σενάριο business as usual, δηλαδή χωρίς να υπάρξουν αλλαγές. Και ε, το ποσό αυτό είναι πολύ μεγάλο για να είναι αληθινό, διότι είναι ε, το διπλάσιο από την αναπτυξιακή βοήθεια που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μία επιπρόσθετη ερώτηση Μπορείτε να κάνετε και ένα προγνωστικό για το σύνολο των εσόδων τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύστημα αυτό. Ε, ήσασταν γενικός, μπορείτε να μας απαντήσετε πιο λεπτομερώς σε αυτό το σημείο. Εμείς έχουμε κάνει υπολογισμούς αυτής της φορολογίας ε, υπολογίζοντας ότι θα μειωθούν οι συναλλαγές ε, και κοιτάζοντας πώς θα ήταν ε, αν υπήρχε κάποια φορολογία κειμενόμενοι. Δηλαδή ε, στα συμβόλαια αγοράς πετρελαίου τα οποία ε, είναι βραχυπρόθεσμα, δηλαδή ε, αγοράζονται και πουλούνται εντός 4 λεπτών. Αυτά θα επιβαρύνονταν με την φορολογία και δεν θα γινόντουσαν πλέον. Αυτός είναι και ο στόχος της φορολογίας, δηλαδή να εξαλείψουμε τους κερδοσκόπους αυτούς από τις αγορές. Εάν σκεφτείτε όμως ότι στην Ευρώπη το, η συνολική παραγωγή ε, ανακυκλώνεται 100 φορές σε ευρωπαϊκές χρηματαγορές ακόμη και αν μειωθούν κατά 60 έως 80% οι συναλλαγές θα παραμείνει μία πολύ σημαντική φορολογική βάση αλλά ομολογώ ότι πρόκειται για προσωμιώσεις δεν είναι προγνωστικά είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει κανείς σοβαρά τα βάραμε ορισμένες προϋποθέσεις ε, αληθοφανές προϋποθέσεις αγοράζοντας μία πραγματική ε, με ε, με μετοχή οπότε τα 5 basis points δεν ε, παίζουν κάποιο μεγάλο ρόλο σε για στις 10.000 ευρώ. Οπότε όσο ισχυρότερη είναι αυτή η φορολογία τόσο αυξάνεται ε, το κόστος της συναλλαγής άρα τόσο θα μειωθούν οι συναλλαγές. Ε, όσο αυξάνουμε ε, τη φορολογία όπως παραδείγματος χάρη όχι για απλές συναλλαγές αλλά για παράγωγα δεν έχουμε όμως ερευνήσει εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνη της εισήγαγε μια τέτοια φορολογία ποιο ποσοστό θα μπορούσε να διαφύγει σε άλλα χρηματοοικονομικά κέντρα. Αλλά λόγω του προβλήματος των ζωνών, δηλαδή δεν μπορεί κανείς να κάνει τις ευρωπαϊκές συναλλαγές ή τουλάχιστον όχι ολικά, μόνο μερικά σε άλλες ε, περιοχές γεωγραφικές. Οπότε ε, δεν νομίζω ότι θα επηρέαζε πάρα πολύ η γεωγραφική παράμετρος το στόχο του προγράμματος αυτού το οποίο σκεφτόμαστε. Εν μέρη απαντήσατε στο τέλος ε, της παρέμβασής σας ένα από που ήθελα να θέσω και που αφορούσε όχι την ε, μετεγκατάσταση σε περίπτωση ε, φόρων ε, ευρωπαϊκών μόνο για τις συναλλαγές, τις σηματοπιστωτικές αλλαγές, αλλά από το Λονδίνο στη Νέα Υόρκη ή στο Χονγκ Κόνγκ. Γιατί οι επιπτώσεις δικτύου ή οι επιπτώσεις εξωτερικότητας, αν είναι σε θέση για να κάνουν αυτή τη μετακίνηση, είναι δυνατόν να γίνει. Η απάντησή σας είναι η... Είναι χρονική η διαφορά της ώρας. Ίσως να έχετε και άλλες απαντήσεις, δεν ξέρω. Αλλά μιλήσατε μόνο για διαφορά της ώρας. Υπάρχουν άλλα επιχειρήματα. Θα ήθελα να γνωρίζω συγκεκριμένα με ποιο μηχανισμό θα μπορούσαμε να το καταπολεμήσουμε. Αν τυχόν γίνει τέτοιο είδους μετακίνηση των συναλλαγών που γίνονται προς μια άλλη ε, χρηματοπιστωτική αγορά. Άρα λοιπόν με ποιο μηχανισμό αν φτιάξουμε αυτό το φορορό στην Ευρώπη θα μπορούσαμε να φορολογήσουμε τις συναλλαγές που γίνονται αλλού αλλά που μας αφορούν. Για παράδειγμα, αν έχουμε ένα παράγωγο προϊόν μιας μεγάλης ε, ευρωπαϊκής πολυεθνικής ε, του πετρελαίου σε μια ευρωπαϊκή αγορά σήμερα και άμα αυτή η πολυεθνική αποφασίσει να φτιάξει αυτό το προϊόν αλλού, το παράγωγο, στην ε, δική της θηγατρική trading. Ποια τεχνικά μέσα μπορούμε να έχουμε για να θεωρήσουμε ότι από τη στιγμή που είναι Ευρωπαίος οικονομικός φορέας θα, φορέας, θα τον φορολογήσουμε. Έπειτα, θα ήθελα να γνωρίζω και ποια είναι η άποψη του Διεθνέου Νομισματικού Ταμείου. Συμμερίζεστε την ανάλυση που γίνεται ή έχετε αντιπιχειρήματα στην ιδέα επιβολή φόρου σε μια ζώνη του κόσμου. Και έπειτα μια άλλη ερώτηση. Αναφέρετε το Μαρόκο αναφέρεται τη Νέα Υόρκη, αλλά δεν αναφέρεται τη Γενέβη. Είναι το ίδιο, έχουμε το ίδιο ωράριο εκεί και υπάρχουν ήδη αγορές χρηματοπιστωτικές εκεί. Νομίζω λοιπόν πως αυτό δεν εμπίπτει στα αντιπιχειρήματα που εσείς ε, προτάξατε. Ähm, Νομίζω ότι όπως και σε θέματα φοροαποφυγής το πολιτικό βάρος της Ευρώπης είναι αρκετά ισχυρό ώστε με απαλές πιέσεις να πείσει την Ελβετία και το Λίχτενστάιν. Δηλαδή, εάν θελήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, εάν λυθεί το πολιτικό θέμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή, εάν αποφασίσει αρχίσει να εισαγάγει μία τέτοια φορολογία στις συναλλαγές δεν νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος των συναλλαγών θα διαφύγει στην Ελβετία. αν φύγουν αυτές οι, ε, οι συναλλαγές, εάν δηλαδή η βραχή ε, πρόθεσμη συναλλαγή δεν λαμβάνει πλέον χώρα στην Ευρώπη, ποιο είναι το πρόβλημά μας, ποιο είναι το μειονέκτημα, κάπου αλλού μπορεί να κάνουν ε, κερδοσκοπία αλλά εμείς θα ξαναβρεθούμε ε, και θα υποφεληθούμε από την, ε, τα προσόντα της Ευρώπης που δεν είναι τα χρηματοοικονομικά. Ίσως ε, η, η Γερμανία παραδείγματος χάρη εδώ και αιώνες έχει επικεντρωθεί εις την πραγματική οικονομία, στη βιομηχανία τα τελευταία 20 χρόνια έχουν γίνει τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και η κερδοσκοπία προϊόντα οικονομικά. Δηλαδή ε, έχει χαθεί ίσως ο στόχος ε, της ταυτότητας με αυτή την ε, δημοσιονομική καπιταλιστική ιδεολογία η οποία δεν μας ταιριάζει τόσο σε εμά τους Ευρωπαίους όσο στην Αμερική διότι η Wall Street είναι εδώ και 150 χρόνια μέρος της βορειοαμερικανικής οικονομικής ε, παιδείας, πράγμα το οποίο δεν ισχύει εδώ. Ε, εδώ μιλάμε απλώς για δεκαετίες και Υπάρχει και, άλλο ένα θέμα. Γιατί δεν μπορούν να μετακινηθούν οι χρηματοοικονομικές συναλλαγές, διότι συνδέονται με προϊόντα. Ένα από τα πιο σημαντικά παράγωγα στη Φραγκφούρτη είναι το DAX Future, που αναφέρεται εις τον δίκτυ των συναλλαγών. Άρα δεν μπορείτε να διαπραγματευτείτε ε, ε, ε, μπορείτε και στις Ηνωμένε Πολιτείε να διαπραγματευτείτε το DAX αλλά όσο, ε, όσο οι μετοχές οι γερμανικές συναλλάσσονται εις την Φραγκφούρτη δεν μπορείτε, να, μπορείτε μεν ε, να έχετε τις, ε, ε, τις συναλλαγές του δίκτυ και στην Αμερική αλλά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα ίσως γιατί τη Γενέβη. Όπως σας είπα, η Ευρώπη ε, και ε, ε, δεν μπορεί η Ελβετία να γίνει μία όαση όπου θα συγκεντρωθούν όλα τα κερδοσκοπικά κεφάλαια αν δεν το επιθυμεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι μία απάντηση, διότι διαφορετικά μπορείτε να γίνετε καζίνο και νομίζω ότι η Ελβετία έχει αντιληφθεί και από από την ισοτιμία του ελβετικού φράγκου και από άλλους παράγοντες ότι εδώ και, ε, ε, και μερικό καιρό ε, βρίσκεται σε μειονοεκτική θέση. Καταρχήν διαφωνώ με τον Στεφάνη για το διαφορετικό ωράριο. Δεν υπάρχει λόγος να μην κάτσεις ξύπνιος, ας πούμε, μια ολόκληρη νύχτα με τέτοιους μισθούς που παίρνει. Αλλά ε, είναι δυνατόν να, να γίνει μερής φορολογία. Ας πούμε, το πρώτο είναι το θέμα της εκαθάρισης. Τι είναι το ευρώ. Είναι το νόμιμο νόμισμα της Ευρωζώνης που είναι μόνο υπάρχει μόνο ως ε, ε, λογαριασμός με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν μπορεί να υπάρξει ε, μια ρύθμιση σε εξωτερική εκτός χωρί, εκτός Ένωσης, εκτός Ευρωζώνης, χωρίς την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Δεν μπορεί να κάνεις συναλλαγή σε λίρες τερλίνες χωρίς την συμμετοχή της Εθνικής Τράπεζας Αγγλίας. Κάθε χώρα πρέπει να το κάνει. Έπειτα έχουμε την ιδέα του ε, του δασμού ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο και ε, Σκεφτείτε την, ολόκληρη την οικονομία να είναι φτιαγμένη σε ένα μόνο νησί. Μετά υπάρχουν οι μετοχές και τα ομόλογα και μετά παράγωγα. Παράγωγα των παραγόντων ο παράγωγα. Ωστόσο θα πρέπει να υπάρχει μια πραγματική οικονομία κάπου και η πραγματική οικονομία είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι η μεγαλύτερη οικονομία. Μπορείτε να πάτε σε παράγωγα τρίτου, τέταρτου επίπεδου, αλλά σε κάποια στιγμή θα πρέπει να υπάρχει και ένα ίχνος αυτών στην πραγματική οικονομία και η ιδέα να φορολογηθούν μονομερώς αυτές οι ε, συναλλαγές ήταν να, να, να συλληφθεί αυτό το ίχνος, να μπορέσουμε να το εντοπίσουμε. Ε, για την περίπτωση του δασμού shares and bonds, etc., you often go and hedge in the spot market. Του, του Βρετανικού φόρου θα είναι με βάση την ε, λίρα. Ε, σε, με βάση το ευρώ θα ήταν η φορολογία που προτείνεται. Άρα λοιπόν η ουσία είναι πως εάν θεωρείτε πως ε, θέλετε να κάνετε μια εφή πολιτική που καταλαβαίνει την αγορά και δεν περιορίζεται σε ένα συγκεκριμένο ποσοστό φορολογίας, αλλά είστε έτοιμος να έχετε ένα ευέλικτο ε, ποσοστό φορολογίας, να δείτε πώς θα λειτουργήσει η αγορά και πώς θα, και πώς θα αντιδράσουν οι διάφορες αγορές, μπορεί να χρησιμοποιήσεις τα εργαλεία που έχει στη θέση του και μπορείς να καλύψεις το 70% του φορολογήσιμου ποσού σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα είχες με μια παγκόσμια ε, συμφωνία. Ακόμα λοιπόν και χωρί παγκόσμια συμφωνία το 70% μπορεί να φορολογηθεί. Επισήμω να σας πω εγώ ότι ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εργάζεται για μια έκθεση για τον G20 ε, και ο κύριο Σούλ συμμετέχει σε αυτή την εκπόνηση αυτή της έκθεσης θα δείτε κάποια πράγματα που δεν χρειάζεται να τα πω ξανά, υπάρχουν στο έγγραφό μου, αλλά ας πούμε τα, τα, τα speed loans αναφέρθηκαν, είναι κάπως επαναστατικό αυτό, υπάρχει και μια πρόσφατη έκθεση για το πώς θα πρέπει να χειριστούμε τις ροές κεφαλαίων και εδώ υπάρχει μια επιτόπου στροφή, ότι δηλαδή στο, στο Διεθνές Ομισματικό Ταμείο, ότι δηλαδή για ορισμένες μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μην πλημμυρίζει δηλαδή τη μια μέρα από ροές κεφαλών και από την άλλη μέρα να υποφέρεις από έλλειψη κεφαλαίων. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι ολοκληρώνεται το πρώτο πάνελ και ερχόμαστε στο δεύτερο πάνελ. Παρακαλώ τους μιλητές να έρθουν εδώ στο Προεδρείο και να καθίσουν. Περνάμε στο δεύτερο πάνελ για θέματα κλιματικών αλλαγών, τον αντίκτυπο της κρίσης στις αναπτυσσόμενες χώρες και το εμπόριο. Να σας παρουσιάσω τους τρεις πανελίστες μας. Εξεβονίμων κάθεται ο κύριος Αμάρ Μπατατσαρίγια, διευθυντής ε, του G24 στη Washington. Πρόκειται για μια ομάδα 24 χωρών από την Αφρική, τη Λατινική Αμερική και την Ασία. Ο δεύτερος προσκεκλημένος είναι ο κύριος Αρουνάμπα Γκος από το Πανεπιστήμιο Πρίστον και η κυρία Νούρια Μολίνα, τη διευθύντρια της Eurodat, του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το Χρέος και την Ανάπτυξη. Ο πρώτος ο κύριος Μπατατσαρίγια. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την μεγάλη μου ευχαρίστηση για τη συμμετοχή σε αυτήν την ακρόαση και τη συμβολή μου στην συζήτηση υπό το πρίσμα των αναπτυσσομένων χωρών. That, uh, the crisis of course showed uh, Καταρχήν ήθελα να πω δύο λόγια ε, για την αποσύνδεση που ήταν όχι μόνο πρώιμη αλλά και άκερη και άσκοπη. Η κρίση μέσω του εμπορίου επηρέασε βαθύτατα τις αναπτυσσόμενες χώρες. Μάλιστα, η πιστοτική κρίση για τις ε, αναπτυσσόμενες χώρες ήταν πολύ πιο δεινή από ό,τι για τις ανεπτυγμένες. Και να μην ξεχνάμε και την εκτόξευση των ε, τιμών πρώτων υλών στα ύψη. Βέβαια, οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι πιο προσάρμοστες, έχουν ισχυρότερους ε, και ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, Βέβαια θα υπάρξουν αναπτυξιακά κενά, θα παραμείνουν και πολλές επιπτώσεις στην παγκόσμια διακυβέρνηση σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά. Σε ό,τι αφορά τον αναπτυσσόμενο κόσμο, είναι τρεις από τις τέσσερις μοχλούς της παγκόσμιας οικονομίας και ανάπτυξης και όπως βλέπετε πριν την κρίση ήταν 80% της ανάπτυξης στον κόσμο που προερχόταν από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Μετά την κρίση και πάλι το 80% της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης θα προέλθει από τον αναπτυσσόμενο κόσμο. Βέβαια, η ιστορία δεν περιορίζεται στην Ινδία, την Κίνα και τη Βραζιλία, είναι πολύ πιο ευρύτερη. Και στις χώρες μέσου οδήματος, από τις 86 ε, χώρες, 67 έχουν ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούσαν τα 4 τα πριν την κρίση και από τις 48 χώρες χαμηλού εισοδήματος 38 ε, έχουν ε, αριθμούς ανάπτυξης και πάλι άνω του 4% και μετά την κρίση. Βέβαια τα αναπτυξιακά χάσματα είναι τεράστια και ο μέσος όρος ε, κατά την ημέρα για τον πλούσιο κόσμο είναι 114 δολάρια και στον ρωτησόμενο κόσμο 1,5 δολάριο ενώ υπάρχουν και σε ορισμένε χώρες στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι κάτω από 10 δολάρια, πολύ πιο κοντά δηλαδή στις χαμηλού εισοδήματος χώρες και στις περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες είναι 3 με 4 δολάρια κατά κεφαλή την ημέρα εισόδημα. 78% των φτωχών ζουν σε αυτές τις χώρες μέσου εισοδήματος. Ακούσαμε για την παγκόσμια διακυβέρνηση και το G20 δεν πρόκειται να μακρηγορήσω για το G20. Θα ήθελα να πω πάντως ότι αυτό που δεν έχει γίνει πλήρως αντιληπτό είναι ότι το G20 έχει μια καλά συγκροτημένη δομή και γερά θεμέλια. Η δομή αυτή καθιστά το G20 μια διαδικασία ένταξης και συμμετοχής, αλλά και αποτελεσματική και μετρήσιμη από ότι το G7. Το G20 δεν έχει γραμματεία, αλλά όπως σας είπα, έχει γερούς δεσμούς με επίσημους θεσμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Παρά την επιτυχία του G20, που μας εξιστόρισε πριν ο κύριος Παντώας Σόπα. Αυτό που μας ενδιαφέρει περισσότερο σήμερα είναι οι προκλήσεις. Θα είναι πιο δύσκολο για το G20 ε, να πραγματοποιήσει κάποια πράγματα στο μέλλον από ό,τι πριν από λίγο καιρό. Ο συντονισμός των στρατηγικών εξόδων από την κρίση θα είναι πιο δύσκολος. Ήδη άρχισε να φαίνεται αυτό. Και η εφαρμογή του πλαισίου είναι πολλά υποσχόμενη μεν, αλλά ας μην υποτιμούμε τις δυσκολίες αυτής της έμπρακτης εφαρμογής. Σε ό,τι αφορά και το νομοθετικό σκέλος, αλλά και την ε, ε, εξέταση από τους ε, ομότιμους εταίρους, να μην το ξεχνούμε, και τις επιρροές της κρίσης στην κλιματική αλλαγή. Αλλά η βαθύτερη κρίση είναι η κρίση της νομιμοποίησης και της συμμετοχής. Όπως είπε ο κύριος Παντόα, ένα τρόπο εξόδου από την κρίση είναι με καλύτερου δεσμού και πιο αποτελεσματικού με του επίσημου θεσμού. Όχι μόνο το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά και με τα Ηνωμένα Έθνη. Το G20 θα πρέπει να συνάψει δεσμού και με τα Ηνωμένα Έθνη και να χρησιμοποιήσει τη μόχλευση σε άτυπε ομάδε, είτε είναι το G24, η Αφρικανική Ένωση, η ΑΣΕΑΝ, η ΠΕΚ και ούτω καθεξής. Βέβαια, έχουμε και την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο, διεθνεί δεσμού. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί μια όθηση όχι μόνο ε, για μια αναθεώρηση της παγκόσμιας διακυβέρνηση μέσω του G20, αλλά επανέφεραν το Διεθνέ Ομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα από τη χώρα των νεκρών. Η κρίση κατέδειξε σημαντικές αδυναμίες στη δομή διαχείρισης αυτών των δύο θεσμών. Και οι αδυναμίες εντοπίστηκαν σε τέσσερα επίπεδα. Υπάρχει ασυμφωνία σε ό,τι αφορά τις βασικές αποστολές των δύο αυτών θεσμών. Οι θεσμοί αυτοί δεν είχαν επαρκείς πόρους για να ανταπεξέλθουν στην αποστολή τους. Τρίτον, υπήρξε διαφωνία ως προς το είδος των μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται για αυτούς τους δύο θεσμούς. Και πρώτα απ' όλα, πάνω απ' όλα, δεν υπήρξε συμφωνία για το πώς θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος διακυβέρνησης για να είναι πιο συμμετοχικός. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες θα βαρύνουν πολύ σε ό,τι αφορά την πρόοδο που θα συζημιωθεί σε θέματα αναθεώρηση παγκόσμια διακυβέρνηση αυτού του δύο θεσμού, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, βέβαια. Είπαμε Είχαμε αρκετά φιλόδοξου στόχου για το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο το 5%, 3% για την Παγκόσμια Τράπεζα. Το θέμα είναι αν θα υπάρξει και πολιτική βούληση για την υλοποίηση αυτών των στόχων. Και αν μιλούμε για μία μάχη στα χαρακόμματα, εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Αν όντω θα υλοποιηθούν οι αλλαγέ που προανήγγυλαν οι G20. Αν δούμε τα σημεία στο Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, Είχαν γίνει κάποιες μεταρρυθμίσεις μέσω της μεταρρύθμισης του Απριλίου 2008 στην Παγκόσμια Τράπεζα και της ε, Τράπεζας Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το σημείο θετηρίας ήταν καλύτερο, αλλά και εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό αν θα υπάρξει υλοποίηση των αλλαγών. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που εμφανίζεται ιδιαίτερα στα πλαίσια της μεταρρύθμισης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Την τελευταία δεκαετία διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία διαρθρωτική μετάβαση άνευ προηγουμένου. Και αν δούμε το μερίδιο των αναπτυσσομένων χωρών στην παγκόσμια οικονομία, μέχρι το 2000 περίπου, η ε, κατάσταση παρέμενα μετάβλητη. Τώρα βέβαια, Βλέποντας τις διαφορές μεταξύ του 2005 και του 2009, διαπιστώνουμε τεράστιες αλλαγές και μεταστροφές. Κάθε χρόνο η μεταβίβαση από τις ε, αναπτυγμένες αναπτυσσόμενες είναι περίπου 100, κάτι που δεν ε, είχαμε διαπιστώσει σε προηγούμενες περιόδους. Να πω δύο λόγια και για την ε, Παγκόσμια Τράπεζα. Η Παγκόσμια Τράπεζα έχει εξίσου σημαντικό ρόλο με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σε ό,τι αφορά την ε, αντίδραση στην κρίση. Δεν έχει τύχει αρκετή προσοχής. Τα τελευταία 15 χρόνια είχαμε 3 εκατομμύρια σε ιδιωτικές ώρες κεφαλαίου προς τον αναπτυσσόμενο κόσμο και αν δείτε την πράσινη γραμμή βλέπετε ότι είχαμε 0 από το σύστημα MDB για την περίοδο αυτή. Και αν θέλετε μία χρηματοπιστωτική αρχιτεκτονική ισχυρή είναι να προσδιοριστεί το σύστημα MTB. Μόνο αυτό θα γίνει όμως αν επιτρέψουμε σε χώρες όπως την Κίνα και την Ινδία να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά τους και για την ανάπτυξη και όχι μόνο για την ανακύκλωση του δημοσιονομικού ελλείμματος στον ΗΠΑ. Αυτά προς το παρόν, τα υπόλοιπα αργότερα. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Αρανάμπ Χαγκός. Thank you, Chairman Klins, and uh, other members of the Special Committee. And... Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, κύριε Ευρωβουλευτέ, σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε να μιλήσω για την παγκόσμια διακυβέρνηση, το κλίμα και το εμπόριο εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης. Το πρώτο που θέλω να πω είναι ότι βασικά έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια πρόκληση παγκόσμιας διακυβέρνησης σε ένα πλαίσιο όπου έχουμε μια πολλαπλή κρίση όπου συγκλίνει ταυτόχρονα οι λύσεις θα χρειαστούν διαφορετικές χρονικές κλίμακες ε, για να επιτευχθούν. Έχουμε τώρα μια οικονομική κρίση όπου η παροδία των πολιτικών είναι γενικά να ζητούν αυξημένη ανάπτυξη και επασχόληση. Επίσης έχουμε τον κίνδυνο αύριο ή μεθαύριο να έχουμε μια αύξηση προστατευτισμού του εμπορίου αν ε, συνεχιστεί η κρίση. Και έπειτα υπάρχει και μια τρίτη απειλή, το... η κλιματική αλλαγή που είναι πολύ πιο μακροπρόθεσμη η κατάσταση. Το θέμα είναι έχουμε τα θεσμικά όργανα, τα μέσα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα ενώ ταυτόχρονα θα διατηρούμε υπόψη μας σε αυτές τις διαφορετικές χρονικές κλίμακες. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε τρεις, τρία σύνολα ερωτήσεων. Πρώτον, πώς επηρεάζει η κρίση την ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές. Δεύτερον, πώς επηρεάζει το πουτυμπόριο, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλος, θα προσπαθήσω να εστιάσω την παρέμβασή μου σε ορισμένες, στην απόδοση ορισμένων κυβερνήσεων βράχη και μέσο πρόθεσμα. Πώς επηρεάζεται καταρχήν η ανταπόκριση στις κλιματικές αλλαγές. τα περιβαλλοντικά ωφέλη της κρίσης κατά κάποιο τρόπο είναι σύντομα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας εκτιμά πως υπήρξε 3% μείωση των εκπομπών το 2009, πράγμα που θα οδηγήσει σε 5% σωρευτικά μείωση μέχρι το 2020. Αλλά δεν πρέπει να είμαστε και τρελά ενθουσιασμένοι περί αυτού, γιατί αυτό που σημαίνει βασικά είναι ότι από τη στιγμή που θα υπάρξει οικονομική ανάκαμψη, οποιοδήποτε είδος ωφέλους ε, μπορεί να ε, διαγραφεί γιατί έχουμε άλλες προκλήσεις για την ανακατανομή των οικονομικών πόρων και μιλάμε βασικά για 11 γιγατόνους ε, αύξηση ε, στις εκπομπές μέχρι το 2020. Το βασικό θέμα που επηρεάζει τις κλιματικές αλλαγές είναι η ανακατανομή των πόρων. Στα πρόσφατα χρόνια, 2004 με 2007, βλέπουμε με αυτό εδώ το γράφημα ότι υπήρξε μια αύξηση στις επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά αυτό άρχισε να πέφτει κάπως. Ε, αυτό σήμανε μια μαζική αύξηση στις δυνατότητες ανανεώσιμης ενέργειας. Ε, μέχρι το 2008, 25% των επιπλέον, ε, της επιπλέον παραγωγής ενέργειας ήταν στον ανανεώσιμο τομέα. Αυτό όμως που έκανε η κρίση είναι οι τριμηνιαίες επενδύσεις αρχίζουν να πέφτουν από τις αρχές του 2008 μέχρι τα μέσα του 2008 και στις αρχές του 2009. Ένας ε, παράγοντας ήταν ε, τα, οι δαπάνες για, τις, για τα κίνητρα, τα πράσινα κίνητρα, που έγιναν, συνολικά καμιά πεντακοσαριά δις δαπανήθηκαν σε, σε 20 χώρες. Εδώ βλέπουμε τι γίνεται στις 20 χώρες του G20. Αλλά βεβαίως υπήρξαν και προκλήσεις όσον αφορά πραγματικά την διάχυση αυτών των κονδυλίων. Η μεγάλη πρόκληση λοιπόν για τη διακυβέρνηση των κλιματικών αλλαγών είναι πώς αντιμετωπίζουμε την προσοχή απέναντι στην προφύλαξη. Δηλαδή πώς πώς καλύπτουμε τα ελλείμματα σήμερα, ενώ ταυτόχρονα προφυλασσόμαστε για τις προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε με το κλιμα... τις κλιματικές αλλαγές. Τι κάνουμε με τις, ε, την αρχιτεκτονική πάνω προς τα κάτω ή κάτω προς τα πάνω και η Κοπεχάγη εδώ ήταν πολύ σημαντική ω προ αυτό. Και έπειτα πώ συνδυάζονται οι μονομερεί δράσει των κρατών από την μια πλευρά με τι πολυμερεί, τι λογικέ δράσει από την άλλη πλευρά. Και έχω την εντύπωση πω θα υπάρξει μια τάση προ το πρώτο, προ τι μονομερεί δράσει δηλαδή. Πράγμα που δημιουργεί πρόβλημα όσον αφορά την ε, πολυμερή και τη διαχείριση των κρίσεων και την ε, παγκόσμια διακυβέρνηση. Τώρα, όσον αφορά τον όγκο εμπορίου, είδαμε τη μεγαλύτερη μείωση του 2009. 12% μεγαλύτερη πτώση μετά από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Ίσως είναι λίγο περίεργο αυτό το γράφημα, ε, να το καταλάβατε, αλλά βασικά εκτός από την Ευρώπη, όπου υπήρξε πολύ μεγάλος αντίκτυπος, η Αφρική, η Μέση Ανατολή και οι χώρες της, ε, της, της Ρωσικής Ομοσπονδίας είχαν τεράστιες μειώσεις ε, τεράστια πτώση στο εμπόριο. Αυτό οδήγησε σε μεγάλες αυξήσεις στην ανεργία. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια ανθρώπους χωρίς δουλειά σε ολόκληρο τον κόσμο. Επίσης ε, έχουν μειωθεί οι αποστολές χρημάτων στις φτωχότερες χώρες. Ε, για ορισμένες χώρες ήταν τεράστιο εισόδημα. Αν έρχεται στο 1 τέταρτο του εθνικού του εισοδήματος ε, τα χρήματα που στέλνουν οι μετανάστες πίσω. Τα εμβάσματα δηλαδή. Ε, η αξία των εξαγών, ας πούμε, για την Αφρική το 2009 έπεσε κατά 32% σε σχέση με το παγκόσμιο μέσο όρο του 33%. Οπότε οι αναπτυσσόμενες χώρες, οι φτωχότερες χώρες, στην ουσία χτυπήθηκαν περισσότερο από την κρίση αυτή ως προσορισμένες επιτυχίες. Επίσης θα πρέπει να θυμόμαστε πως υπάρχει ο κίνδυνος να αυξηθεί ο προστατευτισμός. Μέχρι στιγμής δεν είδαμε σημαντική αύξηση στους εμπορικούς φραγμούς. Εδώ σε αυτό το γράφημα βλέπουμε ότι τους τελευταίους 6 μήνες οι εμπορικοί φραγμοί που εισήχθησαν από τις χώρες G20 και η κάλυψη αυτών των φραγμών για παγκόσμιες εισαγωγές ε, μειώθηκαν. Αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να θυμόμαστε πως δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση και ότι υπάρχει δυνατότητα οι φραγμοί αυτοί να αυξηθούν και το γράφημα αυτό σας δείχνει ότι ενώ οι έρευνες αντι-dumping έχουν ε, μειωθεί, οι, οι έρευνες για ασφαλιστικές δικλείδες στις χώρες G20 έχουν αυξηθεί. Στα τρία λεφτά που μου μένουν θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, στα οποία θα πρέπει να εστιάσουμε βράχη πρόθεσμα. Όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, το πρώτο που θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να διατηρήσουμε τιμέ άνθρακα που μπορεί να κινητοποιήσουν τι επενδύσει. Έχω μιλήσει σε κυβερνήσει, έχω μιλήσει με ιδιώτες επενδυτέ, αλλά με την τιμή αυτή δεν πρόκειται να κινηθούν οι επενδύσεις που θα βοηθήσουν να ξεπεραστεί η κρίση. Δεύτερον, θα πρέπει τα ε, χρήματα για τα πράσινα κίνητρα που δεν έχουν δαπανηθεί δεν θα μετακινηθούν σε άλλους τομείς. Δεν θα μεταφερθούν σε άλλους τομείς. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα γίνουν οι δαπάνες αυτές για πράσινα κίνητρα. Και έπειτα θα πρέπει να είμαστε βέβαιοι ότι η χρηματοδότηση 30 εκατομμυρίων δολαρίων που έχει προβλεφθεί στην Συμφωνία της Κοπεχάγης θα δαπανεθούν. Δηλαδή, Είμαστε ήδη τέσσερις μήνες μέσα στο 2010 και θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο να βρούμε πόρους καθώς και προορισμούς για την δαπάνη αυτών των χρημάτων. Αλλά αν δεν το κάνουμε αυτό θα αυξηθεί η το έλλειμμα που υπάρχει στις ε, διαπραγματεύσεις για το κλίμα. Ταυτόχρονα, μεσοπρόθεσμα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα αυξηθεί το εμπόριο με τις φτωχότερες χώρες. Ακόμα και αν η Βρασιλία και, το, και η Κίνα προσπαθούν και καταφέρουν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα για χώρες όπως ε, χώρες της Αφρικής, ακόμα και μεγάλες τράπεζες χρεώνουν διπλά για την ε, για την χορήγηση πιστώσεων, πράγμα το οποίο ζημιώνει πάρα πολύ τις δυνατότητές τους να συμμετέχουν στο σύστημα. Θα πρέπει να ενισχυθεί δε η διακυβέρνηση και πέρα από την κρίση. <coughs> Για τις κλιματικές αλλαγές θα πρέπει λοιπόν να σκεφτούμε πώς μπορεί να αλλάξει η αρχιτεκτονική του καθεστώτος. Θα μπορούσα από αυτό να σας μιλήσω με περισσότερες λεπτομέρειες κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Αλλά αυτό που φαίνεται να γίνεται είναι ότι εισάγεται περισσότερη ευελεξία στο καθεστώς. Αυτό έχει νόημα μέσα στη μέση μιας κρίσης, αλλά κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, αλλά θα πρέπει να το κάνουμε πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να υπάρξουν εποπτικές δυνατότητες για τις κλιματικές αλλαγές όχι μόνο σε, μονο, σε πολυμερές επίπεδο, αλλά και σε μονομερές επίπεδο. Θα πρέπει να δημιουργηθεί ένας πιο διαφανής μηχανισμός χρηματοδότησης και γι' αυτό θα μπορούσα να μιλήσω κατά τη διάρκεια της συζήτησης και έπειτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε συνδέσεις κλίματος σε όλες τις διαστάσεις, όχι μόνο για τις ε, συνοριακές προσαρμογές, αλλά εκεί όπου γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τις υπηρεσίες και τα αγαθά. Πώς αντιμετωπίζουμε τον προστατευτισμό για τις υπηρεσίες ε, περιβαλλοντικές που προέρχονται από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και τέλος, για το εμπόριο θα πρέπει να εστιάσουμε για στη διακυβέρνηση του εμπορίου και όχι μόνο στο γύρο του, της Δόχα. Θέματα εποπτείας, βελτίωση της διαφάνειας του ΠΟΕ, είναι πολύ σημαντικά αυτά. Βελτίωση πρόσβασης στους μηχανισμούς ε, διευθέτησης κρίσεων, ε, μάλλον διαφωνιών και έπειτα δημιουργία κάποιων δικτύων ασφαλεία για τι πιο ευάλωτες οικονομίε. Όλα αυτά θα ήταν πολύ σημαντικά. Εδώ θα σταθώ λοιπόν και τα υπόλοιπα κατά τη διάρκεια τη συζήτηση. Σα ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Νούρια Μολίνα. Παρακαλώ. Καλησπέρα σα Και πάλι σας ευχαριστώ που μου επιτρέψατε να έρθω. Θα ήθελα να ξεκινήσω με μία γενική σχολίαση του που βρισκόμαστε και αν υπάρχει ανάπαυση ή όχι. Εδώ βλέπετε μία εικόνα του Economist από το 2008 και αντικατοπτρίζει πώς πιστεύαμε πολύ ή τουλάχιστον όσοι ασχολούνται εδώ και πολλά χρόνια για, με την παγκόσμια διακυβέρνηση και τη μεταρρύθμισή της Πώ πώς θα μπορούσαν να βελτιώσουν αυτή την ε, κατάσταση που εξηγείται πάρα πολύ ωραία σε αυτό το, ε, την πρώτη σελίδα του Economist στο εξώφυλλο. Λοιπόν, ε, τώρα σκεφτήκαμε ότι μπορούσαμε να γυρίσουμε πίσω στο 19ο αιώνα διότι το είδος των ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων που χρειαζόμαστε δεν έχουν γίνει ή γίνονται μπαλώματα και όχι ουσιαστικές λύσεις και απαντήσεις και πρέπει αυτό να το σκεφτόμαστε και για να μην χάσουμε την ευκαιρία και να μην χάσουμε ε, την κατεύθυνση την οποία, την οποία θέλουμε να ακολουθήσουμε διότι νομίζω ότι υπήρξε μία πολύ καλή παρουσίαση του τι συμβαίνει στις υποανάπτυξη χώρες οπότε δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία έχουν λεχθεί, αλλά θα ήθελα να σας πω ποιες είναι οι επιπτώσεις ε, της κρίσης που ανάπτυξαν χώρες και ιδίως ε, ε, τις χώρες με χαμηλό επίπεδο. Ναι, μεν έχουν προχωρήσει, διότι ήταν λιγότερο ενταγμένες στο διεθνές σύστημα, αλλά ήταν σαν μία σύγκρουση σε, στο ραλοντή είδαμε γενικότερα ότι ναι μεν οι φτωχοί και οι χώρες άντεξαν καλύτερα αλλά αυτό οφείλωτο ε, στο γεγονός ότι είχαν ε, ε, αποθέματα τα οποία εξαντλούσαν και βλέπετε ότι τώρα δεν υπάρχουν πλέον ούτε αποθέματα ούτε αποταμιεύσεις ούτε δυνατότητα να αντεπεξέλθει κανείς και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό γιατί τις, για τις χώρες με χαμηλό επίπεδο δεν μιλάμε μόνο για κράση διότι ε, όταν, ε, όταν ε, πεινούν οι άνθρωποι δεν σκέπτονται αν υπάρχει κρίση οικονομική ή τι άλλο. Οπότε ε, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για όπου έχουν εξαντληθεί τα αποθέματα και αυτό θα δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση η οποία τους έχει απευθυνθεί. Βλέπετε εδώ ότι οι ανάγκες είναι πολύ υψηλότερες από την εξωτερική χρηματοδότηση η οποία ε, χρειάστηκε ε, το 2009 και θα χρειαστεί το 2010. Έχουν μειωθεί πάρα πολύ οι εξωτερικές ροές χρηματοδότησης ε, και ε, η ιδιωτική η ιδιωτική ε, ροή κεφαλαίων δεν αντιστάθμισε αποτελεσματικά αυτά τα οποία μειώθηκαν. Λοιπόν, βλέπετε ότι γενικώ για τις υποανάπτυξη χώρες ε, υπάρχει εξωτερική χρηματοδότηση αλλά ε, τα δύο τρίτα, δηλαδή η Κίνα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τα υπόλοιπα υπόλοιπα δημιούργησαν ουσιαστικά δάνεια, δηλαδή χρέη. Και ε, ε, ε, είναι προήμιο για μια νέα κρίση. Μετά, ποιος ε, λαμβάνει τα χρήματα. Οι χώρες μεσαίου εισοδήματος που έχουν μόνο ή 2% της αντιδράσεως στην παγκόσμια κρίση. Ναι, μεν αντιπροσωπεύουν το 7% του παγκοσμίου ΑΕΠ, αλλά ε, δεν είναι ε, αυτό ένα σημαντικό ποσοστό. Είναι λιγότερο από ό,τι χρειάζονται. Μία άλλη τάση η οποία θα μπορούσε να είναι ανησυχητική είναι ότι τα χρήματα τα οποία πηγαίνουν σε αυτές τις χώρες, ιδίω αυτές που έχουν χαμηλό εισόδημα, θα στηρίξει ως επτοπλίστων τον ιδιωτικό τομέα και αυτό δεν είναι υποχρεωτικά κακό, αλλά οι ροές ε, οι οικονομικές είναι ε, πάρα πολύ, ε, πάρα πολύ ασταθείς και πρέπει να δούμε πού πρέπει να διατεθούν δημόσιοι πόροι για τις πιο φτωχές χώρες. Ποιες είναι λοιπόν οι επιπτώσεις αυτών των αντιδράσεων στην κρίση. Καταρχήν, η ροή προς τις υποανάπτυξη χώρες και τις χώρες χαμηλού εισοδήματος έχουν μειωθεί σημαντικά και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ε, υποκατασταθεί, ε, έχει υποκαταστήσει ε, άλλες χρηματοδοτήσεις και θα έχει μεγάλη ε, σημασία για τα επόμενα τρία χρόνια. Επίσης, το είδος των, της χρηματοδοτήσεως που δίνεται υπό χρέους ουσιαστικά προϋποθέτει ότι θα αποδυναμώσει τη χρηματοδότηση του κράτους και θα μειώσει τη δυνατότητα των χωρών αυτών να αναπτυχθούν καλύτερα και ε, να ε, δημιουργήσουν ε, πολιτικές που θα τους καταστήσουν πιο ανθεκτικές στις επόμενες κρίσεις. Γι' αυτό και είναι σημαντικό ίσως να σκεφτούμε τις υποανάπτυξη χώρες σε δύο επίπεδα καταρχήν για τις πολιτικές οι οποίες σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις χώρες αυτές να γίνουν πιο ανθεκτικές, λιγότερο βάλωτες ε, στα μελλοντικ... στους στις μελλοντικές δονήσεις και ε, τι μπορεί να γίνει χωρίς να επαναλάβουν τις ροές τις οποίες ανάφεραν προλαλήσαντες. Όσον αφορά τις πολιτικές για τις υποανάπτυξη χώρες, εγώ πρέπει να επανέλθω στο ρόλο των διεθνών ε, χρηματοοικονομικών ε, οργανώσεων. Διότι αν μιλάμε για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο καθορίζει υπό ποιου όρους οι οικονομίες αυτών των χωρών ε, θα πρέπει να εφαρμόσουν φορολογικές μακροοικονομικές πολιτικές να μπορέσουν να δανειστούν και από αυτής της πλευράς. Η κοινωνία των πολιτών, η πανεπιστημιακή έχουν κατακρίνει τον τρόπο με τον οποίο ε, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ε, συμβουλεύσει τις χώρες αυτές να απελευθερώσουν και να ιδιωτικοποιήσουν το δημόσιο τομέα, να αλλάξουν ε, φορολογική πολιτική και αυτά ήταν παράμετροι στην, στην κρίση που απεδείχθηκαν ότι δεν ήταν οι καλύτερες μέθοδοι για τις χώρες αυτές. Και τι γίνεται τώρα. Και εδώ ε, διαφωνώ με τον κύριο Βαντσέλμ, ο οποίος έφυγε δυστυχώς από την αίθουσα, αλλά αναθεωρήσαμε ε, τις, ε, τα τελευταία δάνεια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου προς τις χώρες χαμηλού εισοδήματος, οι οποίες δεν, έχουν, δεν δείχνουν να αποκλίνουν από την παλιά πρακτική. Δηλαδή υπάρχει ίσως λίγο μεγαλύτερη ευελιξία διαφορολογική, αλλά όχι πολλά πράγματα. Ε, αυτά τα οποία ελέγχθησαν για το, την οικονομική πολιτική και τον ρόλο ελέγχου του κεφαλαίου ε, ναι μεν είναι θετικά αλλά δεν επιτυχάνουν αυτό που είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Επίσης πέραν από το επίπεδο χώρας ή συγκεκριμένου κράτους, ο κύριος Βαντσέλντ ίσως θα μου έλεγε αν ήταν στην αίθουσα ότι ναι, υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία και ιδίως για την φορολογική πολιτική, αυτό θα βοηθούσε τις χώρες αυτές, αλλά τι θα γίνει όταν θα εξαντληθούν οι πόροι, διότι αναπτύσσουν όλο και μεγαλύτερα δάνεια και χρέη, όπου χρειάζεται πιο γενικευμένη αντιμετώπιση. Ναι μεν το, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ασχοληθεί με τα ελλείμματα, τη μείωση των ελλημάτων αλλά όχι με την αύξηση των εισοδημάτων. Να, μειώνονται, να μειωθεί η φορολογία, να δοθούν φορολογικά κίνητρα σε εταιρείε οι οποίες θα εγκατασταθούν στις χώρες αυτές. Κοιτάζοντας λοιπόν τον ισολογισμό και από τις δύο πλευρές, ναι μεν είναι πολύ σωστό να καταπολεμηθεί η ε, διαφυγή ε, ε, είναι ένα βασικό θέμα για να μπορέσει κανείς να αυξήσει το εσωτερικό κεφάλαιο αλλά ε, ε, δεν μπορεί δεν πρέπει οι πολυεθνικές εταιρείες να ε, δηλώνουν τι κερδίζουν στις χώρες χαμηλού εισοδήματος και εκεί να πληρώνουν το υψηλότερο φόρο πρώτης βαθμίδας. Ε, ότι ουσιαστικά θα έπρεπε να βοηθήσουν τις, ε, αυτές τις χώρες χαμηλών εισοδημάτων. Υπάρχουν και άλλα θέματα πολύ σημαντικά, το ανέφερε ο πρώτος ομιλητής και μετά στη συνέχεια ξαναεπανελήφθη, Δηλαδή, ελέγχθη ότι είναι αναγκαίο να υπάρξει ένα διεθνές νόμισμα, ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούμε να επιλύσουμε ε, ε, ε, να αντεπεξέλθουμε των, ε, των αξιών της στασιμότητος η οποία έχει δημιουργηθεί διότι η, ε, τα δάνεια αυτά είναι πολύ υψηλότερα και κοστίζουν πολύ περισσότερο στις χώρες χαμηλού εισοδήματος από το ποσό το οποίο τους έχει διατεθεί και θα ήθελα να αναφερθώ εις τις μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα και ιδιαίτερο στο Διεθνές Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και τέλος να αναφερθώ στον τρόπο με τον οποίο οι χώρες αυτές αντιμετωπίζουν τα χρέη τους διότι θα πρέπει να υπάρξουν αξίες ενεργητικού που θα τους επιτρέπουν να εφαρμόσουν πολιτικές οι οποίες θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν και να καταρτήσουν πολιτικές για δια διαρκή και δίκαιη ανάπτυξη. Ε, και εκεί θα πρέπει να περιληφθεί ένα άλλο βασικό σύστημα το οποίο αναφέρθηκε, ε, δηλαδή ένας μηχανισμός που θα επιτρέπει να επεμβαίνει κανείς σε μελλοντικές ε, κρίσεις χρεών, ώστε να υπάρχει καλύτερος τρόπος αντιδράσεως. Ευχαριστώ. Και τώρα ερχόμαστε στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων. Η Περβόνς έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ για τις ομιλίες σας. Θα σας παρουσιάσω χίδιν τις ερωτήσεις μου και όποιος θεωρεί ότι είναι κατάλληλο σας απαντήσει. Ως προς τις αναπτυσσόμενες χώρες, συμφωνούμε για το πώς έχουν πληγεί από την κρίση. Διαπιστώνουμε ότι ο κύκλος της ΔΟΧΑ ξεκίνησε στραβά. Όλες οι εμπορικές διαπραγματεύσεις ήταν χρονοβόρες, αλλά ειδικά ο κύκλος της ΔΟΧΑ χρόνισε. Και σίγουρα η χρηματοπιστωτική κρίση δεν διευκόλυνσε την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων. Σίγουρα οι αναπτυσσόμενες χώρες ε, απέφχονται μια πολιτική προστατευτισμού των ε, αναπτυγμένων χωρών. Άρα η Ινδία για παράδειγμα, τι συμφέρον έχει για το πλήσιμο των διαπραγματεύσεων δεδομένου του, των ε, συνεπειών που θα έχει η Ντόχα για τον γεωργικό πληθυσμό της Ινδίας για παράδειγμα. Κάτι που είπα και στο πρώτο πάνελ και αφορά τις ανησυχίες μας για τις κλιματικές αλλαγές και την ανάπτυξη. Είδαμε τα αποτελέσματα της Κοπεχάγης, δεν ήταν και πολύ εντυπωσιακά, στον ΠΟΕ το ίδιο και για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέμε προχωρούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν σας ζητώ καμία θαυματουργή λύση, αλλά προς ποια κατεύθυνση να ψάξουμε. Γιατί στις συνομιλίες με τον Πασκάλ Λαμή μας έλεγε ότι στην Κοπεχάγη όλοι είναι ίση, αλλά δεν υπάρχουν πολλές ελπίδες γιατί δεν υπάρχει συμφωνία. Σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να στραφούμε για να βρούμε κάποια στοιχεία διαιτησίας στην παγκόσμια διακυβέρνηση. Πιστεύετε ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο απομακρύνθηκε από, το, από τη Συμφωνία της Ουάσιγκτον ή στις δράσεις του φαίνεται ότι εμένει σε αυτήν. Κυρία Μολίνα, όλα όσα είπατε για τους λογιστικούς κανόνες και ποια είναι τα αποτελέσματά τους, ώστε οι χώρες να μπορούν να φορολογούν ε, στο έδαφος τους ε, τα έσοδα από τις ε, πρώτες ύλε για να μην υπάρχει διαφυγή φορολογικών εσόδων αλλά συζητώντας με εκπροσώπους αναπτυγμένων χωρών, λαμβάνω την ίδια απάντηση, ότι οι επιχειρήσεις φταίνε. Πιστεύετε ότι είναι αποτελεσματική αυτή η προσέγγιση. Και αν χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αρεσιμότητα για τα δάνεια αυτά και τις προϋποθέσεις για το δανεισμό αυτών των χωρών, σε ποιο επίπεδο θα πρέπει να γίνει. Ε, ας αρχίσουμε με την κυρία πρώτα και μετά με τους άλλους δύο ομιλητές. Για την αιρεσιμότητα θα μπορούσα να κάνω δεκάωρες ομιλίες για κάθε σας ερώτηση, αλλά δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Αυτή ήταν μία από τις προτάσεις ε, που έκανα προς το τέλος της ομιλίας μου. Πιστεύω ότι οι όροι του δανεισμού μεταξύ βορείων και νοτιών χωρών θα... δεν θα πρέπει να στηρίζεται στην ερεσιμότητα των τελευταίων 30 ετών. Την παραδοσιακή ερεσιμότητα της συμφωνίας, ε, της ομοφωνίας του, της Washington αλλά σε κοινά συμφωνημένους κανόνες δανεισμού και λήψης δανείων. Και επίσης χρειαζόμαστε κάποιους ε, κανόνες προφύλαξης, να μην ε, κατασπαταλούνται τα δάνεια, αλλά να χρησιμοποιούνται για τους ε, στόχους που ζητήθηκαν. Αλλά κάτι τέτοιο προϋποθέτει όρους πολιτικής, οικονομικής πολιτικής και μακροοικονομικής πολιτικής. Για πολλούς και διάφορους λόγους, ο πιο σημαντικός όμως είναι ότι και μάλιστα εδώ πιστεύω συμφωνούμε όλοι, και οι μακροοικονομικές συμβουλές που έδωσαν οι βόρειες χώρες προς τον Νότο ήταν εσφαλμένες ως προς την οικονομική πολιτική. Και η προσέγγιση αυτή ήταν λάθος και για, για τον αναπτυγμένο κόσμο, αλλά πολύ περισσότερο για τον αναπτυσσόμενο. Ο εκπρόσωπο του διεθνού Νομισματικού Ταμείου είπε ότι δίνουμε στον καθένα τι συμβουλέ που πιστεύουμε ότι χρειάζεται. Οι αναπτυσσόμενε χώρε όμω δεν χρειάζονται η ίδια μακροοικονομική πολιτική ή δημοσιονομική πολιτική, η πολιτική χρέους σαν αυτή που χρειαζόμαστε εμεί ο αναπτυγμένο κόσμο. Και τέλος, υπήρξε ενδιαφέρον για απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση πολλών κλάδων στι αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν θα αποκαλέσω αυτή την προσέγγιση συνομωτική, αλλά σίγουρα εξυπηρέτησε ορισμένα εμπορικά συμφέροντα των βόρειων χωρών. Η ιδιωτικοποίηση του χρηματοπιστωτικού κλάδου άφησε ανοιχτά διάπλατα τι πόρτες για τράπεζε των ε, βορείων τραπεζών. Και αυτό ε, αύξησε την πληκτικότητα, την ταυλιτότητα της κρίσης. Η κρίση πάντως ε, μας δίνει την ευκαιρία να διδαχθούμε από τα παθήματά μας και να δούμε πού έσφαλαν όλες αυτές οι μακροοικονομικές πολιτικές. Ίσως ο βαθμός ε, κεφαλαϊκής διαχείρισης ε, ή αποτελεσματικών βιομηχανικών πολιτικών, ο έλεγχος των χρηματοπιστωτικών ροών, γιατί όχι, και των εμπορικών ροών. Και ο προστατευτισμός δεν είναι πάντα κακός για μια χώρα χαμηλού εισοδήματο. Για την πρώτη σας ερώτηση. Και την πρώτη σα ερώτηση για το τι στάση κατά Γενέβη. Εγώ δεν είμαι διαπραγματευτή τη Ινδία στη Γενέβη, αλλά Πιστεύω ότι θα πρέπει να σκεφτούμε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Το πρώτο είναι τα εμπορικά συμφέροντα των χωρών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και το άλλο, η άλλη πτυχή είναι το πώς λειτουργεί το καθεστώς. Αν σκεφτούμε μόνο τα εμπορικά συμφέροντα, μπορεί να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι στο μέσο μιας κρίσης η Ινδία, η ΙΠΑ, ΕΕ, η Ευρώπη, καθένας προσπαθεί να προστατευτεί. Αλλά βλέπετε ταυτόχρονα πως διαπραγματεύονται σε άλλα φόρα. Ας πούμε, η εμπορική συμφωνία διαπραγματεύεται η Ινδία με την Ευρώπη που μπορεί να υπογραφεί φέτος. Δηλαδή, το θέμα δεν είναι κατά πόσο τα εμπορικά συμφέροντα επικρατούν ή όχι, είναι πού θα επιληθούν αυτά, σε ποιο φόρουμ. Αυτό που ήταν ενθαρρυντικό για μένα ήταν ότι για τη διάρκεια της τελευταίας υπουργική ε, συνεδρίασης που έγινε τον ε, Δεκέμβριο του 2009, διάφορες χώρες, Ινδία, ΗΠΑ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Κίνα, με πολύ διαφορετικά συμφέροντα, Βραζιλία, στο εμπορικό σύστημα, υπέβαλαν κοινή πρόταση για την εξέταση τη λειτουργία και τη αποτελεσματικότητα του εμπορικού καθεστώτο, συστήματο. Αυτό ήταν πολύ ενθαρρυντικό γιατί είναι η πρώτη φορά που αναγνωρίζεται πω κάτι λείπει στη διακυβέρνηση. Και αυτό ακριβώ λέω, να εστιάσουμε όχι μόνο στη διαπραγματεύσει αλλά στην διακυβέρνηση. Και όταν ε, γίνεται, δίνεται έμφαση στη διακυβέρνηση, θα σκεφτούμε πολύ πιο στεναρό ε, μηχανισμό εποπτείας, αύξηση πρόσβασης στην διευθέτηση των ε, διαφορών αν μπουν μέσα και τα συνδεθούν και τα περιβαλλοντικά θέματα, μπορεί να γίνει πιο, πιο περίπλοκος ο μηχανισμός διεθέτησης των ε, διαφορών. Το άλλο θέμα, δηλαδή, πού θα βρούμε τα στοιχεία διακυβέρνησης, είναι πολύ ευρύτερο. Δεν νομίζω πως υπάρχει ένα μόνο πρότυπο το οποίο να μπορούμε να το επιλέξουμε. Αυτό που θα πρέπει να εξετάσουμε είναι ένα σύνολο ερωτήματων, ένα σύνολο θεμάτων. Στα έγγραφά σας υπάρχουν διάφορα ενημερωτικά σημειώματα. Θα πρέπει δηλαδή καταρχήν να δούμε σε ποιο φόρουμ θα αντιμετωπίσουμε τις κλιματικές αλλαγές. Αυτό που έκανε η Κοπενχαουαγή ήταν να προτείνει πως η αρχιτεκτονική από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή στόχων και χρονοδιαγραμμάτων, δεν κατάφερε να μας προχωρήσει πολύ και δεν κατάφερε να ενώσει και τις χώρες που, τις πιο σημαντικές. Λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε και πιο ευέλικτε αρχιτεκτονικέ, όπου οι χώρε θα δίνουν τα δικά του προγράμματα. Ναι, όλα αυτά εντάξει όσον αφορά την ε, πολιτική ε, διεκπαιρέωση. Αλλά από την άλλη πλευρά, με βάση τι τα κρίνουμε όλα αυτά, σε τι βασίζουμε τον επόμενο γύρο διαπραγματεύσεων. Με τι, συγκρίνουμε τα αποτελέσματα και την απόδοσή μας. Βασιζόμαστε σε διμερείς συμφωνίες. Αν αυτές ε, εφαρμοστούν και στις κλιματικές αλλαγές, ε, αν ε, αποκλείσουμε ένα σύνολο φτωχών χωρών θα λειτουργήσει το σύστημα. Δηλαδή αν τα, τα μαγειρέψουν μεταξύ τους η ΙΠΑ, η Κίνα, η Βραζιλία και η Ένωση, ας πούμε, μετά με ρωτήσετε πού θα πρέπει να κατευθυνθούμε. Και εκεί δεν νομίζω πως υπάρχει ένα μόνο πρότυπο. Πρέπει να σκεφτούμε την κλίμακα της χρηματοδότησης, αλλά κανένας από τους μηχανισμούς διακυβέρνησης αυτή τη στιγμή δεν αντιμετωπίζει αυτή την κλίμακα, δεν προβλέπει τέτοια κλίμακα χρηματοδότηση. Επίση, ευελιξία στον τρόπο χρηματοδότηση, δηλαδή σε ποιον δίνει ε, ε, δωρεάν ε, τα χρήματα, σε ποιον δίνει ε, τα soft Πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο μείγμα όλων αυτών. Τα θέματα διαφάνειας και λήψη αποφάσεων για την κατανομή των πόρων, των κονδυλίων. Και τρίτο σημαντικό θέμα για μένα είναι η αξιοπιστία της δέσμευσης, δηλαδή πώς παρακολουθείς τις δεσμεύσεις και πώς διασφαλίσεις ότι θα υπάρχει συμμόρφωση. Η Κοπενχάγη είπε, έκανε κάποιες τέτοιες προτάσεις, αλλά υπάρχουν πολλά ανεπίλητα ζητήματα ακόμα. Πώς θα φτάσουμε στο ανωτοτόριο, ποιο είδους πληροφορίες χρειαζόμαστε, ποιες... Ε, πώς δημιουργείται ένας μηχανισμός εποπτείας από τους εταίρους που να λειτουργεί, δηλαδή δεν είναι απλά οι αναπτυσσόμενες χώρες που εξετάζουν τις εκπομπές ε, των αναπτυγμένων και τούμπαλιν. Ξέρω, ξέρω μακρηγορώ, αλλά ζητώ συγγνώμη αλλά είναι δύσκολο να βρεθούν οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα. Uh, conditionality, you, you... Πολύ σύντομα. Η αιρεσιμότητα ίσως μπορεί να αναφερθεί σε δύο τύπους. Ένα, η συνένεση ε, της Washington ε, το δεύτερο είναι οι κοινωνικές επιταγές στις οποίες όλοι πιστεύουμε αλλά θα τις καθορίσει η Washington ή η χώρα. Και το τρίτο το οποίο είναι πολύ σημαντικό είναι η, η, η ερεσιμότητα της διακυβέρνησης. Ποιος πρόκειται αυτό να το καθορίσει, οι δημοκρατικές διαδικασίες ή η Washington. Όσον αφορά το δημοσιονομικό τομέα υπάρχουν ουσιαστικά δύο βασικοί στόχοι αυτή τη στιγμή. Ο ένας στόχος είναι πώς οι G20 θα νομιμοποιηθούν και θα καταστούν ε, αποτελεσματικοί και δεύτερον ε, είναι το θέμα των δημοσιονομικών οργανώσεων. Πώς θα γίνει πιο αποτελεσματικό ο θεσμός των G20. Θα σας ε, έλεγα ότι από το 1999 ε, έχοντας παρακολουθήσει σαν ε, παρατηρητής αυτές τις συνεδριάσεις μπορώ να σας πω ότι υπάρχει το ερώτημα είναι αν το G20 μπορεί να είναι μια πιο αποτελεσματική διαδικασία. Η απάντηση είναι βεβαίως ναι και ό,τι γίνει στο επόμενο ένα-δύο χρόνια θα έχει πολύ μακροπρόθεσμες επιπτώσεις. Δεύτερον, και εδώ απαντώ στο ερώτημά σας κύριε Πρόεδρε, θα ήταν χειρότερα εάν ε, ε, ε, με τα προβλήματα αυτά χωρίς το G20 παρόλες αυτές τις φυγόκεντρους δυνάμεις ε, που υπάρχουν. Η απάντηση είναι ναι, διότι η G20 ακόμη και στις προτάσεις Ομπάμα όπως ονομάζονται είναι μία δύναμη η οποία επαναφέρει τους ενδιαφερόμενους στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όπως είπαμε είναι μία δύναμη η οποία ε, επιτρέπει να υπάρχει ε, ε, απολογισμός και τρίτον χρειάζεται μεγαλύτερη φιλοδοξία, πρέπει να αλλάξουμε το μοντέλο και την διακυβέρνηση και όλα αυτά είναι στενά συνδεδεμένα. Θα σας δώσω το παράδειγμα της παγκόσμιου τραπέζης. Στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής της, κάθε, ε, κάθε Υπουργό ο οποίος παρενέβη ε, είχε αμφιβολίες εάν η Παγκόσμια Τράπεζα χρειάζεται χρηματοδότηση. Όλοι είπαν ότι χρειαζόμαστε, θα χρειαστούμε μεγαλύτερη Παγκόσμιο Τράπεζα μετά από αυτή την ε, ε, κρίση, άρα θα χρειαστεί να χρηματοδοτήσουμε την τράπεζα αυτή. Γιατί, διότι υπάρχουν διαφορετικές φωνές, διαφορετικές ψήφοι. Λέγω λοιπόν ότι αν δεν θέλετε να ε, χρησιμοποιήσετε τα χρήματά σας εμείς μπορούμε να καλύψουμε μεγάλο ποσοστό, μεγαλύτερο ποσοστό αλλά να έχετε υπόψη σας ότι αυτό θα έχει επιπτώσει στη διακυβέρνηση δηλαδή δημιουργούνται νέες ευθύνε. Σαν Ευρωπαίοι λοιπόν σας καλώ να πείτε ότι εάν έχουμε περισσότερο, ε, πιο ισχυρή φωνή θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε με τους οργανισμούς. Έχω και εγώ μερικές ερωτήσεις, για να είμαι κάπως προκλητικός. Δεν θα έπρεπε να έχουμε και μια παγκόσμια χρηματοπιστωτική οργάνωση, όπως έχουμε μια παγκόσμια οργάνωση εμπορίου, για να θεσπίζει προδιαγραφές, να έχει δικαίωμα επιτήρησης και να διαθέτει και μηχανισμό επιβολής κυρώσεων και όσοι θέλουν να είναι μέλη αυτής της οργάνωσης να δέχονται και τους κανόνες συμμετοχής. Δεύτερον, οι αναπτυσσόμενες χώρες υποφέρουν όλες από παραοικονομία, από φοροδιαφυγή και από σχετικά υψηλή διαφθορά όχι στο ίδιο επίπεδο όλες οι χώρες, αλλά όλοι υποφέρουν από αυτά τα τρία δεινά. Και όταν μιλούμε για πακέτα διάσωσης και αναπτυξιακή βοήθεια, δεν ασχολούμαστε με συστηματικό τρόπο με αυτές τις τρεις μάστιγες των αναπτυσσομένων χωρών. Η κυρία Μολίνα είπε να μην αποκλίνουμε από την ορθοδοξία, από το ορθοδόγμα. Εγώ νομίζω ότι μετά την κρίση από πολλούς τρόπους αποκλίναμε από το κύριο, από το κρατών δόγμα. Ακόμη και η Ευρωπαϊκή Ένωση φαίνεται ότι αποκλίνει από τον σωστό δρόμο όπως τον κρίναμε. Εγώ είμαι φιλελεύθερος και πριν από τρία χρόνια δεν θα συμφωνούσα με προτάσεις που σήμερα επικροτώ. Άλλο ερώτημα ο ρόλος της Κίνας και της Αφρικής. Ποιος θα είναι. Και ο Πασκάλ Καμφά έχει κάποιες ερωτήσεις, γι' αυτό στη θέση τώρα για να ολοκληρώσουμε. Είχαμε πάει πριν από λίγους μήνες με κάποια μέλη της Επιτροπής σε συνάντηση με το Συμβούλιο του ILO και πρότειναν ε, να συνταχθούμε καλύτερα με τις απαιτήσει πολιτικής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Γιατί λοιπόν να μην γίνει μια σύμπραξη στις αναπτυσσόμενες χώρες μεταξύ Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και Διεθνούς Γραφείου Εργασίας. Γιατί υπάρχει τραπεζική πτυχή, αλλά υπάρχει και κοινωνική πτυχή. Και εκεί θα μπορούσαν να αλλάξουν οι προδιαγραφέ πολιτική που προτείνει σήμερα το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο, αν υπήρχε μια καλύτερη συνεργασία με την Διεθνή Οργάνωση Εργασία. Σε ό,τι αφορά τι κλιματικέ αλλαγέ. Τι γνώμη έχετε για την πρόταση σε ό,τι αφορά ένα φόρο προστιθέμενη αξία του άνθρακα, κάτι αντίστοιχο με το ΦΠΑ για τον άνθρακα, ώστε να τιμολογείται διαφορετικά ο άθρακα σε διάφορες περιοχές του κόσμου, χωρίς να διαταράσσονται όμως συνθήκες ε, θεμητού ανταγωνισμού. Ποια είναι η γνώμη σας. Με την ίδια σειρά παρακαλώ απαντήστε. Για την ε, συγκεκριμένη ερώτηση κοινών αποστολών ε, του Διεθνούς Ομισματικού Ταμείου με άλλες οργανώσεις όπως η Παγκόσμια Οργάνωση Εργασίας έγιναν κάποια τέτοια πειράματα στην Ουκρανία. Και είναι χρήσιμε τέτοιε συνεργασίε γιατί προσθέτουν και άλλε προοπτικέ. Ένα από τα διαφορετικά προβλήματα του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου είναι ότι δεν ιδρύθηκε για, για οικονομία αναπτυξιακή. Δεν έχει αναπτυξιακούς οικονομολόγους, ούτε σχεδιάστηκε για να αντιμετωπίσει να βοηθήσει χώρε χαμηλού εισοδήματος. Και υπήρξε μία παρέκκληση από την αρχική εντολή του Διεθνούς Ομεσματικού Τάμιου προκειμένου να ασχοληθεί αυτό και με τις χαμηλές, ε, χαμηλού εισοδήματος χώρες. Γι' αυτό και είναι και μικρής εμβέλεια τέτοιου είδου συμπράξει. Σε ό,τι αφορά το, τη χρηματοδότηση από τις χώρες του Βορρά προς τον Νότο. Γιατί όχι. είπατε ότι ως φιλελεύθερος θα ήσταν πιο απρόθυμος ως προς την καινοτομία από το ορθόδογμα. Ίσως για λόγους παγκόσμιας διακυβέρνησης δεν χρειάζεται, σαν και καλά δημιουργούμε νέα, νέους θεσμούς. Και υπάρχουν και κάποιες προδιαγραφές για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας. Σχολείται και το ΩΣΑ, κάποια σώματα του ΟΗΕ καλό θα ήταν να αξιοποιήσουμε καλύτερα τις ισχύουσες, τι υπάρχουσε δομέ. Ίσως δεν υπάρχει μια, ανάγκη μια νέα οργάνωση παγκόσμια παγκόσμιο οργάνωση δωρητών, αλλά καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχουσών δομών. Αυτέ οι προδιαγραφέ είναι αντικείμενο συμφωνία μετά από μια διαπραγματευτική διαδικασία που θεωρείται νομότυπη και από τι δύο συμβαλόμενε πλευρέ γιατί μερικές φορές ο τρόπος διαχείρισης της ε, βοήθειας δεν κρίθηκε ούτε νομιμοποιημένος, ούτε ισορροπημένος, ούτε θεμητός. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει ισορροπημένη εκπροσώπηση τέτοιου είδου διαπραγματεύσει μεταξύ Βορρά και Νότου, ώστε πραγματικά το αποτέλεσμα είναι αντικείμενο συμφωνία. Σε ό,τι αφορά την απόκληση από το κρατών δόγμα. Νομίζω ότι αυτό χρειαζόμαστε, να αποκλίνουμε από το ορθοδόγμα, όχι να εμείνουμε εκεί. Ενώ αυτό που βλέπουμε είναι μια αιμονή στο δόγμα. Ο, τελευταίο ο τελευταίος ομιλητής από το προηγούμενο πάνελ είπε ότι εμείς στην Ευρώπη δεν έχουμε παράδοση χρήσης οικονομιών κερδοσκοπικών δραστηριοτήτων. Και ότι κερδίζουμε τα χρήματά μας με την παραγωγή βιομηχανικών αγαθών. Οπότε τέτοιου είδου αναπτυξιακές στρατηγικέ και βιομηχανικέ πολιτικέ που ακολουθήσαμε είναι αυτέ που δεν επιτρέψαμε τα τελευταία 30 χρόνια στις αναπτυσσόμενες χώρες. Γι' αυτό και εδώ χρειαζόμαστε μια αλλαγή πορείας. Πολύ γρήγορα, μία ερώτηση θα προσπαθήσω να απαντήσω. Το θέμα του φόρου προστιθέμενης αξίας άνθρακα. Προτιμώ έναν φόρο άνθρακα από ότι ένα παγκόσμιο συντονισμένο σύστημα εμπορίας άνθρακα, γιατί κάτι τέτοιο προϋποθέτει επιδόματα κατανομής, κάτι που προϋποθέτει κίνδυνο και διαφθοράς, ανάγκη καλύτερης επιτήρησης. Είναι πολύ πιο περίπλοκος ο συντονισμός παγκοσμίω τέτοιων συναλλαγών και εμπορίας. Βέβαια, ο ΦΠΑ άνθρακα δημιουργεί πολλές επιφυλάξεις και ερωτηματικά. Για παράδειγμα, η Κίνα, που, που γίνεται ο μεγαλύτερο ρηπαντή ε, αυτή τη στιγμή με διοξίδιο του άνθρακα, είναι όχι επειδή θέλει να εκπέμπει διοξίδιο του άνθρακα, αλλά επειδή είναι το μεγαλύτερο πλέον εργοστάσιο στον κόσμο η Κίνα. Οπότε σίγουρα θα υπάρξει επιρροή στη μεταπληκτική βιομηχανία της ε, Κίνας και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα της διαφυγής ε, του άνθρακα με τη μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων και να δούμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητας σε μεμονωμένους κλάδους. Ένα άλλο μείζον ζήτημα είναι πώς θα γίνει ο συντονισμό μεταξύ των διαφόρων δικαιοδοσιών. Μονομερό βέβαια μπορεί κανεί να επιβάλλει άνθρακα στην επικράτεια, φόρο άνθρακα στην επικράτειά του, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα, η δυνατότητα μάλλον, και έχουν υποβληθεί σχετικές προτάσεις, το διεθνέ Νομισματικό Ταμείο να γίνει φόρουμ για το συντονισμό του επίπεδου τη φορολογία. Και ένας άλλος προβληματισμός που ανακύπτει είναι αν τα έσοδα αυτά που συγκεντρώνονται σε μία δικαιοδοσία θα παραμείνουν εκεί ή θα ιδρυθεί ένα παγκόσμιο ταμείο που θα συγκεντρώνει όλα αυτά τα έσοδα από ένα τέτοιο φόρο. Και ίσως μια πρόταση συνδυασμένη, μεικτή, ένα τμήμα των πόρων να δρομολογείται προς αναπτυσσόμενες χώρες. σε έναν ρυθμισμένο κόσμο υπάρχει μακρο και μακροπρονοητική διάσταση που είναι του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι μακροδιαστάσεις δεν περιλαμβάνει μόνο τις τράπεζες αλλά και τις ασφάλειες, ε, την αγορά των χρεογράφων, λογιστικά, καθεστώτα για την αφαιρεγκαιότητα, εταιρική διακυβέρνηση. Οπότε Όλα αυτά αντιμετωπίζονται στο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τώρα. Και η διακυβέρνηση αυτού του Συμβουλίου έχει γίνει ουσιαστικά ένα G20, γιατί είναι ίδιοι. Είτε μας αρέσει είτε όχι, έτσι έχουν τα πράγματα σήμερα. Και ίσως είναι και καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Δεν πιστεύω ότι θα ήταν εύκολο να δημιουργήσουμε μια παγκόσμια οργάνωση χρηματοπιστωτικών συναλλαγών που θα είναι υπεροργάνωση. Σε ό,τι αφορά την παραοικονομία και τη διαφθορά, είναι τεράστιο πρόβλημα. Αλλά η κινητοποίηση, η εσωτερική η χώρα κινητοποίηση πόρων σε, όλο, σε όλες τις αναπτυσσόμενες χώρες έχει αυξηθεί εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία. Στην Ινδία, για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή είναι 35 με 40% του ΑΕΠ. Στην Λατινική Αμερική έχει αυξηθεί κατά 30%, το ίδιο και στην Αφρική. Οπότε κάτι κάνουν σωστό αυτές οι αναπτυσσόμενες χώρες, παρόλο που μπορεί να θέλει να κάνουν και περισσότερα. Τώρα, απόκληση από το ορθό δόγμα. Πολύ μου άρεσαν αυτά τα λόγια, γιατί γι' αυτό παραπονιόμασταν πριν την κρίση, ότι για τις αναπτυσσόμενες χώρες υπήρξε πλήρης απόκληση στις αναπτυσσόμενες ε, χώρες, αλλά εμονή στις αναπτυγμένες χώρες για λόγους που ήταν είτε άλλες φορές καλοί και άλλες φορές κακοί. Για την Κίνα και την Αφρική. Υπάρχει περισσότερη συμπληρωματικότητα στο ρόλο της Κίνας, της Ινδίας και άλλων ε, ε, παραγόντων κατά των ε, χωρών ΔΑΚ. Εκεί το 80% της βοήθειας στόχο έχει τη στήριξη του κοινωνικού τομέα και του προπολογισμού. Για την ε, Κίνα, την Ινδία και τις αραβικές χώρες, το 80% των χρημάτων πηγαίνουν στην υποδομή και άρα τη χρηματοδότηση των δανείων. Η Κίνα, η Ινδία και οι αραβικές χώρες χρηματοδοτούν μια μισή φορά περισσότερο τις υποδομές της Αφρικής ενώ η Παγκόσμια Τράπεζα, η, από την Παγκόσμια Τράπεζα την ε, ε, Αφρικανική Τράπεζα Ανάπτυξη και όλες τις υπόλοιπου δωρητές μαζί. Η ενεργειακή ικανότητα της Αφρικής θα εξαπλασιαστεί. Οπότε χρειάζεται η συμπληρωματικότητα. Αλλά θέλουμε και διαφάνεια και λογοδοσία και δημοσιότητα. Ευχαριστώ, Περβάς. Θέλεις να ανακεφαλαιώσεις. Ευχαριστώ. Όπως συμβαίνει συνήθως αυτές ε, τις ε, ακροάσεις, ε, προσπαθούμε να κάνουμε ε, μία σύνθεση και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Από αυτά λοιπόν που ακούσαμε, ξεκινώντας από τον πρώτο μιλητή μας, ο οποίος ήταν και ουσιαστικός, ε, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συνέλθει από την κατάστασή της, αντί να είναι το θύμα της κρίσεως, θα είναι το θύμα της εξόδου από την κρίση κρίση. Και απαντώντας ένα από τα ερωτήματά σας κύριε Πρόεδρε πρέπει ίσως να αναθεωρήσουμε τον τρόπο με τον οποίο επεμβαίνουμε και διαχειριζόμαστε την εξωτερική μας δράση και νομίζω ότι αυτό για την έκθεση θα είναι πολύ σημαντικό διότι αυτό που ελέγχθη σχετικά με την αποτυχία της μεθόδου συντονισμού και την ε, ε, καλή επίδοση επιτόπου νομίζω ότι συμπληρώθηκε με ε, ε, τα σχόλια που αντάλλαξα με τον κύριο Ότμαρ Κάρας. Οπότε, όσον αφορά την ουσία ε, για μας η ευρωπαϊκή δράση είναι κάτι το οποίο πρέπει να σκεφτούμε διαφορετικά από ό,τι σκεφτήκαμε τη στρατηγική της Λισαβόνας όσον αφορά την ε, περιφερειακή και διεθνή ολοκλήρωση δεν πρέπει ε, όλα να γίνουν συνενετικά για να προχωρήσουμε και αυτό πρέπει να μας έχει γίνει μάθημα διότι εκ του παραλίλου μας παραπέμπει σε αυτά τα οποία είχαμε και στο παρελθόν. Δεν περιμέναμε να ολοκληρώσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, για να κάνουμε διευρύνσεις και αυτό θα κάνουμε και και στο μέλλον. Εάν λοιπόν να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τους, τις συνεργασίες με τους γείτονές με Ελβετίας και άλλους δεν θα έχουμε λύσει ακόμη όλα μας τα προβλήματα. Όσον αφορά το διεθνές νομισματικό θέμα, ότι υπάρχει μία διαστροφή σε ένα σύστημα όπου το διεθνές ε, ε, νόμισμα απόθεμα είναι ε, το νόμισμα μίας χώρας το οποίο δημιουργεί ανισότητες και αποδυναμώνει το, το οικοδόμημα του συστήματος. Επανέρχομαι εις την σχέση μεταξύ νομίσματος και εμπορίου θα πρέπει λοιπόν ε, ίσως να δημιουργηθεί ε, ένας ε, διεθνής νομισματικός οργανισμός οπότε ίσως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα πρέπει να αναθεωρήσει την θέση του και γι' αυτό θα ήθελα να σας πω ότι όσον αφορά το δεύτερο πάνελ το οποίο είχαμε η ιδέα που ότι η Ευρώπη έχει μεγάλη ευθύνη όσον αφορά την παγκόσμια διακυβέρνηση ε, συμφωνώ με τον κύριο Σουμάχερ σχετικά με ε, τα καζίνα στην Αμερική όπου υπάρχουν δίκτυα και στοιχεία δράσης όπου ίσως ε, η ε, αλλαγή γεωγραφικής, ε, γεωγραφικού χρόνου εφόσον και ο τζόγος είναι χρηματονομισματική ενέργεια, είναι πολύ σωστό να συγκρίνεται όσον αφορά τον καπιταλισμό, όπως ε, τον γνωρίσαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και ιδίως ε, στην αρχή είχαμε 30 καλά έτη και μετά έναν καπιταλισμό με στοιχεία ε, επί των οποίων όμως θα έπρεπε να έχουμε οικοδομήσει. Στο, για το τελευταίο πάνελ Σχετικά με το τελευταίο πάνελ, αυτό το οποίο ε, διατηρώ είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει ίδια διακυβέρνηση σε όλους τους τομείς της παγκοσμίου διακυβέρνησης, ακόμη και αν υπάρχουν επαναλαμβανόμενα προβλήματα νομιμοποίησης, αποτελεσματικότητα και ε, ε, αντιπροσωπευτικότητος. Αυτά είναι τα τρία στοιχεία που πρέπει να διατηρήσουμε. Για το G20 νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία ότι το G20 είναι καλύτερο από το G7 αλλά δεν είναι και το τέλειο. Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια διακυβέρνηση ε, καλύτερα οργανωμένη και άρα επανερχόμαστε στο θέμα το οποίο δεν απαντήσαμε όταν ε, συζητήσαμε τα G. Δηλαδή επειδή υπάρχουν G, δηλαδή groups, δηλαδή ομάδες παντού, δεν σημαίνει ότι λύσαμε όλα μας τα προβλήματα και σαν Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Όσον αφορά τις υποανάπτυξη χώρες, η ευθύνη σε σχέση με τους όρους δανεισμού κατά τη γνώμη μου αναφέρεται στον ιδιωτικό και τον δημόσιο δανεισμό και γι' αυτό νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει επίσης να περιληφθεί στην έκθεσή μας γιατί η ε, κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων, μία έκφραση η οποία χρησιμοποιήθηκε από τις πολυεθνικές για να καλύψουν τις επενδύσεις τους υποανάπτυξη χώρες, δεν θα πρέπει να μας ε, ε, καθησυχάσει. Διότι είδαμε ότι οι καλές επιχειρήσεις στις υποανάπτυξη χώρες χώρες είχαν ε, λιγότερα θετικά αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ όπως και όλους όσοι συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια. Σε ευχαριστώ Περβόνς και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους πάντες και τους μιλητές του δεύτερου πάνελ για την υπομονή τους και για την αντοχή τους να παραμείνουν μέχρι τέλους. Ευχαριστώ.